Bonjour euh, tout le monde. Καλημέρα σας. Αγαπητή Βερονίκ, θα περάσουμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα πρέπει να σας πω ότι προτείνουμε κάποιες μικρές αλλαγές και θα πρέπει όπως σας ανακοινώθηκε και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος της Γραμματείας την Παρασκευή να ανταλλάξουμε τα τρία τελευταία σημεία της ημερήσιας διάταξης αύριο για πρακτικούς λόγους. Από τις 4.30 μέχρι τις 5 θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τις βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα. Από τις 5 έως τις 6 θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο και το πάνελ υψηλού επίπεδου για τις χρηματοοικονομικές ροές από την Αφρική. Και από 6 μέχρι 6 και μισή τέλος θα ολοκληρώσουμε με το σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου για την 69η Σύνοδο της ε, Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν εντάσεις ε, για την ημερήσια διάταξη ως τροποποιήθηκε. Όχι. Ωραία, εγκρίνεται λοιπόν. Και να περάσουμε τώρα στα πρακτικά της ε, συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου του 2013. Θα τα λάβατε αυτά. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις, θα πρέπει να τις γνωστοποιήσετε στη γραμματεία πριν το πέρας της συνεδρίασης σήμερα το απόγευμα. Επίσης, θα λάβατε και τις ε, αποφάσεις και τις συστάσεις της συνεδρίασης των συντονιστών της 21ης Ιανουαρίου του 2014. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ε, σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών, θα πρέπει και αυτά να τα επισημάνετε στη γραμματεία πριν το τέλος της ε, ε σημερινής συνεδρίασης. Α, ιδάλλως θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται αυτές οι αποφάσεις. Είχα προβλέψει επίσης να σας κάνω και μια ανακοίνωση για το Αφγανιστάν αλλά θα το συζητήσω διαζώσεις με τη Βερονίκα αργότερα. Δεν υπάρχουν αιτήματα για ανακοινώσει από τις Επιτροπής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι όμως το οποίο θα θέλετε να μας πείτε. Χωρίς μικρόφωνο η πρόσωπο της Κομισιόν. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε επίση λάβει και ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σημερινή συνεδρίαση. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο σημείο επί της ουσίας στην ημερήσια διάταξη. Η παρουσίαση μιας έκθεσης ε, την οποία ζήτησε η Επιτροπή Ανάπτυξης για το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού στη Δυτική Όχθη από πλευράς ε, διεθνούς δικαίου. Η μελέτη αυτή για αυτό το ευαίσθητο ζήτημα θα μας παρουσιαστεί από δύο εκπροσώπους του Κέντρου Μελετών Διακονά, ένα κέντρο διεθνών μελετών σπουδών και σήμερα έχουμε δύο εκπροσώπους, την κυρία Μάλιν Γκρίνχιλ και τον κύριο Ζάκουτ. Θα δώσω απευθείας το λόγο λοιπόν στους εκπροσώπους της ε, Διακονά και νομίζω ότι η κυρία Γκρίνχιλ είναι αυτή η οποία θα λάβει πρώτη το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μας που μας έχετε προσκαλέσει σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε τη νομική ανάλυση για τον χωροταξικό σχεδιασμό του τομέα C της Δυτικής Όχθης και να δούμε και την συμμετοχή στην ανάπτυξη της περιοχής. Από ιδεολογική και ιστορική σκοπιά έχει γίνει περιγραφή τη διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη και γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τα δικαιώματα και τον έλεγχο τη γη. Και όλα αυτά εμπίπτουν ε, στο διεθνές ε, ε, δίκαιο, στο κρατος δικαίου, σε περίπτωση που υπάρξει δυνατότητα ανάλυσης και πραγματικής επίλυσης της κρίσης. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η δυτική όχθη είναι υποκατοχή. Βάσει συνήθους διεθνούς δικαίου, μια περιοχή θεωρείται υποκατοχή όταν είναι υπό την εξουσία ενός εχθρικού στρατού. Το διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο στη γνωμοδοτήσή του που έκανε το 2004 επιβεβαίωσε ότι η Δυτική Όχθη, μεταξύ της οποία, στην οποία περιλαμβάνεται και η Ανατολική ε, ε, Ιερουσαλήμ και η Λωρίδα της Γάζας, και εδώ θα ήθελα να σας παραθέσω, να τα πω λίγο πιο αργά, μάλιστα. Ναι, ναι, θα μιλάω πιο αργά. Um, so, in the International Court of Justice... Στη γνωμοδότηση λοιπόν του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου του 2004 επιβεβαιώθηκε ότι η Δυτική Όχθη που περιλαμβάνει και την ε, Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζης αποτελεί κατεχόμενη περιοχή και το Ισραήλ είναι η ε, κατοχική δύναμη. Βάσει διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, της νομοθεσίας που αφορά τον πόλεμο λοιπόν και τα ανθρωπιστικά δικαιώματα, ε, όλα αυτά ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. Κάτι το οποίο έχει επαναληφθεί επανειλημμένως με διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου των Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης. Επομένως υπάρχει πρόβλεψη μεταξύ άλλων για την ευημερία του Παλαιστινιακού λαού. Η παρουσίαση αυτή επικεντρώνεται στη δράση της κατοχικής δύναμης, αλλά δεν θα πρέπει να αρνούμαστε ότι υπάρχουν και ε, αντίστοιχες ε, ένοπλες ε, πράξεις και από την Παλαιστινιακή Αρχή. Βάσει της Σύμβασης της Γενέβης ε, θα πρέπει να υπάρχει πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλα τα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη προστασία όταν υπάρχει ε, σύραξη. Υπάρχουν ε, κατευθυντήριες γραμμές τη Ευρωπαϊκής Ένωση για τη συμμόρφωση με το ανθρωπιστικό δίκαιο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την τήρηση αυτής της νομική υποχρέωσης. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση εξαρτάται φυσικά και από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται όλα αυτά τα στοιχεία. Το κέντρο Διάκονα, το οποίο εκπροσωπούμε, έχει ως στόχο να δώσει αντικειμενική και στρατηγική ανάλυση για το διεθνές δίκαιο. Μία από τις πρόσφατες εκθέσεις μας είναι η νομική ανάλυση του χωροταξικού σχεδιασμού που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Δυτική Όχθη. Το καθεστώς αυτό ε, είναι στον πυρήνα της όλης διαδικασίας επικισμού. Ελέγχονται άνω του 60% των εδαφών της Δυτικής Όχθης. Εδώ είναι οι διάφορες περιοχές που αναφέρονται στις συμφωνίες του Όσλο και ο χωροταξικός σχεδιασμός αποφασίζει ποιος κατασκευάζει τι και πότε. Ε, υπάρχει έλεγχος φυσικών πόρων, ε, θαλάσσιες οδοί, υδάτα και ούτω καθεξής ε, και φυσικά θα πρέπει να καθορίζεται και σε ποιο βαθμό μπορούν να αναπτυχθούν οι παλαιστινιακές κοινότητες. Ο τομέα C έχει ανατεθεί από τις Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και ε, αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ε, φιλοδοξία βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους ε, υποσκάπτεται από την όλη διαδικασία. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει καμία ελπίδα λύσης δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου του 2012 για την προαγωγή της Παλαιστινιακής Ανάπτυξης μέσω μιας διαδικασίας η οποία προβλέπει και συμμετοχή της τοπικής Παλαιστινιακής κοινότητας αλλά και Ισραηλινών. Θα ήθελα επίσης να σας παρουσιάσω... Συγγνώμη, πρέπει να μιλάσετε πιο αργά, μας διαβάζετε, δεν μας μιλάτε και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας μεταφράσουν οι διερμηνείς. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω πόσο σημαντικό είναι ο χωροταξικός ε, σχεδιασμός στον τομέα C. Έχουμε δύο χάρτες, ένα από το Συντονιστικό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και σε αυτό το χάρτη βλέπετε ότι ο τομέας C είναι ε, ο τομέας ο οποίος είναι σκιασμένος με μπλε χρόνια, χρώμα. Περιλαμβάνει πάνω από το 60% της δυτικής όχθης και αυτό είναι το ουσιαστικό, είναι υποκατοχή και ο Ισραηλινός στρατός ε, έχει τον έλεγχο και τον, ε, από πλευράς ασφαλείας και από πλευράς διοικητικού ελέγχου. Περιλαμβάνεται τους περισσότερους από τους φυσικούς πόρους, πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, καθώς επίσης και αρρώσιμη γη. Ο τομέας αυτός έχει περιορισμούς για τους Παλαιστινίους και για τον τομέα C και για όσους διαμένουν στον τομέα Α και Β. Και εδώ είναι τα μόνα εξωτερικά σύνορα που έχει η Παλαιστίνη πέραν ε, των σύνορων με το Ισραήλ και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το εμπόριο. Ο περιορισμός που, θα, ε, που έχετε εδώ, τα όρια δηλαδή, περιλαμβάνει και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι για ε, επικισμό. Τα πιο σκούρα χρώματα είναι οι επικισμοί που έχουμε στη δυτική όχθη. Στα δεξιά σας έχετε τους επικισμούς και από την άλλη έχουμε τους φυσικούς πόρους, ε, συγγνώμη, στα αριστερά είναι οι επικισμοί και στα δεξιά είναι ο χάρτης με τους φυσικούς πόρους και κάτω, στον κάτω χάρτη έχουμε τις στρατιωτικές περιοχές. Όλες αυτές οι περιοχές είναι πολύ σημαντικές για την άμεση αλλά και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κατεχόμενης περιοχής και όπως σας είπα και προηγουμένως και τη βιωσιμότητα οποιοδήποτε μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. με εξαίρεση την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ο υπόλοιπο τομέα ΣΕΙ είναι αυτό ο οποίο περιλαμβάνει του επικισμού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ του, ε, της περιοχή του τομέα ΣΕΙ, που όπω καθορίζεται στι συμφωνίε του Όσλο, και την ε, περιοχή η οποία έχει Ισραηλινού επικισμού. Εδώ τώρα έχετε αυτό το χάρτη. Λυπάμαι πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν τα βλέπετε και πολύ καλά. Ο οποίο δείχνει που υπάρχουν επικισμοί και ποιες περιοχές έχουν ε, ε, καθοριστεί για επέκταση των επικισμών. Επίσης, στο χάρτη αυτό θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι μπλε κύκλοι και αυτοί οι μπλε κύκλοι δείχνουν τι κατεδαφίσεις έχουν γίνει και τι εκτοπισμοί γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις και ε, βλέπετε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στις περιοχές των επικισμών. Οι περιοχές οι οποίες σημειώνονται με αστερίσκο είναι οι περιοχές τις οποίες έχουν εκτοπιστεί οι Παλαιστινιακοί πληθυσμοί. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε διάφορες δομές οι οποίες έχουν κατεδαφιστεί και άνθρωποι οι οποίοι εκτοπίστηκαν από το 2009 στο 2013 με αριθμητικά στοιχεία πλέον. Ε, το σκούρο είναι οι κατεδαφισμένες ε, εκτάσεις και το μπλε ε, πλαίσιο είναι οι εκτοπισμένοι. Και εδώ βλέπετε ότι είναι ανωδική η τάση Για το 2013 έχουμε στοιχεία μέχρι τον Αύγουστο. Ο εκτοπισμός αυτός ε, και οι κατεδαφίσεις είναι ε, συνεχώς σε αύξηση από τότε που συνάφθησαν οι συμφωνίες του Όσλο και όλα αυτά ε, διέπονται και από το χωροταξικό σχεδιασμό στον τομέα C. Συνειδητοποιούμε βέβαια ότι όλα αυτά δεν είναι και κάτι καινούριο, ότι οι προκλήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού είναι πολύ σημαντικές. Ο συνάδελφος θα σας τα αναφέρει ε, εντό ολίγου. Είναι πράγματα τα οποία γνωρίζει η Επιτροπή σας και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπάρχει και μία έκθεση από το 2011 η οποία λέγεται «Χωροταξικό σχεδιασμό του τομέα C» και εκεί ε, λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και της Παλαιστινιακής κοινότητας και θα πρέπει να υπάρχει και λογοδοσία για την βοήθεια που δίνεται στον τομέα C και φυσικά να υπάρχει και σημαντική αύξηση της βοήθειας. Υπάρχει και ένα ψήφισμα από τον Απρίλιο του 2013 και στο ψήφισμα αυτό, όπως επίσης και στο πρόγραμμα δράσης για τη Δυτική Άχθη, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν συνάδει με το διεθνές ε, δίκαιο στον τομέα C. Τι πρέπει να γίνει τώρα. Θα πρέπει να ε, δούμε πώς μπορεί να γίνει η συμμέρφωση με αυτές τις ε, πολιτικές. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να μελετήσουμε αυτό το χωροταξικό σχεδιασμό. Αξιολογούμε με τα νομικά αίτια τα οποία χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να χρησιμοποιήσει αυτό το χωροταξικό σχεδιασμό και αξιολογούμε και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις παλαιστινιακές κοινότητες και την, ε, τα συνέπεια στην ανάπτυξη αντιστοίχως, καθώς επίσης και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του καθεστώτος αυτού και του μηχανισμού που ε, χρησιμοποιείται για να υπάρξει ο χωροταξικός ενδιασμός. Ολοκληρώνουμε με κάποιες συστάσεις και με κάποια συμπεράσματα προς όλους τους ενδιαφερομένους, ε, συμπεριλαμβανομένους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ένωσης. Ο συνάδελφος τώρα θα σας δώσει κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το χωροταξικό σχεδιασμό και το κατά πόσον είναι νόμιμο. Παρακαλώ. Παρακαλώ συνεχίστε. Εάν μπορούσατε να μας μιλάτε θα είναι πιο απλό και για την ε, μετάφραση. Ευχαριστώ. Ως σημείο αφετηρίας πρέπει να πω ότι υπάρχει διαρκής ε, διαφιλονικία για τα θέματα του χωροταξικού σχεδιασμού και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και το ίδιο για το διεθνές δίκαιο που διέπει τις δραστηριότητε αυτές, σε περιπτώσει κατοχής ιδίως. Όμως, ε, επί τη ουσία, μιλάμε για προβλήματα βραχυπρόθεσμα περισσότερο παρά μακροπρόθεσμα. Να το εξηγήσω. Η ανθρωπιστική βοήθεια, ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων και οι διάφορες καταδαφίσεις διασυνδέονται με την επέκταση των, ε, των επικισμών. Τώρα, εάν ο χωροταξικός σχεδιασμός ε, με τη στρατιωτική κατοχή της Δυτικής Όχθης έχει οδηγήσει σε παράνομες δράσεις που αντιφάσκουν με το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό χρειάστηκε να προβλέψουμε ε, τις εξηγήσεις, να χρησιμοποιήσουμε τις εξηγήσεις που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινές αρχές για να παρέμβουν στον χωροταξικό σχεδιασμό. Και γι' αυτό ανατρέξαμε στο διεθνές νομικό πλαίσιο που απαγορεύει την παρέμβαση της δύναμης κατοχής κατά τη δίκηση των κατεχόμενων εδαφών και των πληθυσμών που κατοικούν εκεί. Έτσι μπορέσαμε να αναλύσουμε το νόμιμο του χωροταξικού σχεδιασμού, των αρχών και των πρακτικών που ακολουθήθηκαν, όπως ε, υλοποιήθηκαν στην, στον τομέα ΣΥ. Μιλάω αρκετά... Ε, απλά <laughs> υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Όχι, υπάρχει το πρόβλημα, διαβάζετε. Η διοίκηση των ε, κατεχόμενων εδαφών σε κάθε περίπτωση κατοχής σημαίνει ότι αυτοί που δικούν τα κατεχόμενα εδάφη θα πρέπει να δρουν προς όφελος όλων των πληθυσμών που εκεί κατοικούν. Το διεθνές δίκαιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διατηρεί το status quo όταν υπάρχει κατοχή σε εξέλιξη κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η προσάρτηση επιπλέον εδαφών με τη χρήση βίας. Αυτό απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Σε καιρούς κατοχής, ωστόσο, υπάρχουν κάποια απαγορευτικά όρια, όπου η δύναμη κατοχής μπορεί να ε, παραβεί με δική της νομοθεσία ή δικούς της νόμους. Πολλές φορές αυτού του είδους οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ως σκοπό την ε, ομαλή εξέλιξη της ζωής των πολιτών ή την λειτουργία μιας νόμιμης κυβέρνησης την ε, πραγματική ασφάλεια των δυνάμεων της δύναμης κατοχής ή τέλο πάντων την ε, κάλυψη των υποχρεώσεων προκύπτουν από τη Χάρτα των Διεθνών ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στο χωροταξικό σχεδιασμό η προέλευση της παρέμβασης είναι στατιστικής φύσεως. με τον νόμο 1971, 618 του 1971. Εκεί τροποποιήθηκε ο νόμος που ήδη υπήρχε για τις δυνάμεις κατοχής προκειμένου να οργανωθούν οι ανάγκες χωροταξικού σχεδιασμού. Στα αριστερά βλέπετε τους νόμους της Ιορδανίας, ενώ βλέπετε από την άλλη τις αλλαγές που πρότεινε η Σέλινη για η δύναμη κατοχής. Ένα σύστημα ολιστικό σφαιρικό δηλαδή, με μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, με συγκεκριμένες επιτροπές χωροταξικού σχεδιασμού που είχαν ε, επιτόπια προγράμματα και μετά με ακόμη μικρότερες τοπικές ε, επιτροπές που φρόντισαν να σχεδιάσουν στην πράξη τον επικισμό οι Παλαιστίνοι είχαν δικαίωμα ε, ιδιοκτησίας πολύ περιορισμένου σε όλη τη διάρκεια αυτής της κατοχής. Μετά από τα χρόνια κατοχής ε, της Δυτικής Όχθης, με το νόμο 418 καταργήθηκαν όλες οι τοπικές επιτροπές που ίσχυαν προηγουμένως για το χωροταξικό σχεδιασμό και ο στρατικός, ο που ήταν ο κεφαλής των δυνάμεων κατοχής ανέλαβε όλες τις αρμοδιότητες αυτών των επιτροπών και δημιούργησε ανάλογα με τη χρονιά τουλάχιστον 20 ειδικέ επιτροπές τους οποίους παρακολουθούσαν οι Ισραηλινές αρχές και οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής με σκοπό ακριβώς να επεκταθούν ε, οι εγκαταστάσεις επικισμού στις περιοχές της Δυτικής Όχθης. Με αυτή τη διαδικασία οι Παλαιστίνοι έχασαν κάθε ε, διάσταση ιδιοκτησίας στην χωροταξία και στο χωροταξικό σχεδιασμό των εδαφών τους. Έτσι, με αυτή την ανάλυση καταλήξαμε στο εξή συμπέρασμα η παρέμβαση στην τοπική νομοθεσία δεν συνείδε με τις υποχρεώσεις της δύναμης κατοχής να συμμορφωθούν με τους τοπικούς νόμους. και χρησιμοποίησαν μια από τις δυνατότητες εξαίρεσης με την πρόβλεψη νέας νομοθεσίας. Ταυτόχρονα, η στετιωτική ε, τάξη, έδωσε στις Ισραηλινές αρχές, στον Ισραηλινό στρατό, ε, διαταγές ε, προκειμένου να ξεκινήσουν πολιτές και, πολιτικές και πρακτικές με μακροπρόθεσμες συνέπειες που αντιφάσκουν με τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στην έκθεσή μας λοιπόν συμπεραίνουμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός στον τομέα C ε, ήταν αντίθετος με τις επιταγές της διεθνούς νομοθεσίας. Η έκθεση καταλήγει και στο εξής συμπέρασμα, ότι υπάρχουν παράνομες πρακτικές ή πολιτικές που εφαρμόστηκαν και διευκολύνθηκαν, εξυπηρετήθηκαν από τα θεσμικά όργανα της ομάδας ορταξικού διαδιασμού των Ισραηλινών. Ένα παράδειγμα. η καταστροφή εγκαταστάσεων ε, της, πολι... ζωής των πολιτών των Παλαιστινίων με σχολεία, λόγω χάρη που καταστράφηκαν, αυτά έχουν καταγραφεί ως εγκλήματα πολέμου και οδήγησαν και στον εκτοπισμό των συγκεκριμένων κοινοτήτων που εξυπηρετούνταν από αυτές τις εγκαταστάσεις, από αυτές τις υποδομές. Όπως επίσης ξύνθηκε ο κίνδυνος εκτοπισμού και πέραν αυτών υπήρχαν συνεχείς δημεύσεις και η παρεμπόδιση της προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό έγινε με μέσα και έτσι παρεμποδίστηκε και η ενίσχυση από την Ευρώπη. Η οικοδόμηση του τείχους και το καθεστώς παρακολούθηση, ελέγχου δηλαδή, προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ με τον διαχωρισμό του υπολείπου της Δυτικής Όχθης, με ένα τέτοιο πρόγραμμα χωροταξικού σχεδιασμού οδήγησε στην ιδιοποίηση εδαφών για την επέκταση των ε, ε, δραστηριοτήτων οικοδόμησης εγκαταστάσεων επικισμού. Οι δραστηριότητες των Ισραηλινών οδήγησαν στην άρνηση του 94% των ε, αδειών ε, κατάσταση των Παλαιστινίων. Μόνο το 1% του τομέα C έχει διατεθεί στην ε, ανάπτυξη υποδομών από τους Παλαιστινίους. Έτσι το 2010 εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος των περιορισμών από τους Ισραηλινούς έφτασε τα 4,05 δις δολάρια. Και σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η συνολική προστιθέμενη αξία από την άρση των σημερινών περιορισμών και την πρόσβαση σε δραστηριότητες και την παραγωγή στον τομέα C μπορεί να φτάνει τα 3,4 δις δολάρια ή 35% του Παλαιστινιακού ΑΕΠ το 2011. Τέλος του παραθέματος. Η διοίκηση των Ισραηλινών κατά τη διάρκεια αυτής της κατοχής έχει οδηγήσει σε μια εξάρτηση των Παλαιστινίων και την, ε, τον περιορισμό του χωροταξικού του σχεδιασμού. Έτσι η μόνη ανάγκη που πραγματικά τους έμενε ήταν η ε, λήψη ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε καιρούς στρατιωτική κατοχής, προφανώς η δύναμη κατοχής έχει την πρωταρχική υποχρέωση να ασχολείται με το, με την επιβίωση και την ε, τις βασικές ανάγκες του κατεχόμενου πληθυσμού. Εφόσον αυτές δεν καλύπτονται, έχει το καθήκον η αρχή κατοχής να επιτρέψει να διευκολύνει την παροχή βοήθειας από τρίτα μέρη. Στην πράξη, όταν ε, μιλάμε για την παροχή βοήθειας, αντιμετωπίσαμε παρόμοια προβλήματα από τους ε, φορείς της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας το ίδιο που αντιμετωπίσαμε όταν οι Ισραηλινοί παρενέβησαν στο Παλαιστινιακό χωροταξικό σχεδιασμό. Λόγου χάρη την καταστροφή ανθρωπιστικών προγραμμάτων και εξοπλισμού, τις κατασχέσεις και δημεύσεις και την παρενόχληση των ε, εργαζομένων στους ανθρωπιστικές οργανώσεις. Και αυτό με στρατιωτικές ενέργειες των δυνάμεων κατοχής. Αυτό οδήγησε στο εξής καταστροφή τουλάχιστον 246 υποδομών που είχαν χρηματοδοτήσει δωρητές από το 2011. Από το 2012 όμως και το 2013 φτάσαμε σε ένα συνολικό κόστος 750 εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία τελικά δεν πέτυχε το στόχο της. Ε, υποδομές που καταστράφηκαν δηλαδή ή ε, ε διαταγές που δεν εκτελέστηκαν. Η κατάσταση αυτή ή τέλο πάντων αυτό το νομικό κενό οδήγησε τι ανθρωπιστικέ οργανώσει να προσπαθούν να βρουν κάποια ισορροπία μεταξύ των επιταγών τη προσφορά ανθρωπιστική βοήθεια και το, το, το κατά πόσον σε περίπτωση μη προσφοράς βοήθειας υπήρχε ε, σχέση με παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η ECRC πρόσφατα αποφάσισε να πάυσει την προσφορά ε, της ανθρωπιστικής της βοήθειας λόγω των παραβιάσεων των Ισραηλινών ε, δυνάμεων κατοχής. Η απόφαση αυτή άρχισε να ισχύει μάλιστα από την περασμένη εβδομάδα. Σημειώνει μάλιστα η οργάνωση αυτή. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι Ισραηλινές στατιωτικές αρχές συνεχίζουν τις παράνομες δραστηριότητέ τους, καταστροφής, ιδιωτική ιδιοκτησίας, του προστατευόμενου κατά τα άλλα πληθυσμού των Παλαιστινίων και είναι απρόθυμες να ανταποκριθούν στις ανάγκες το πληθυσμό αυτού που θα πρέπει να προστατεύεται. Και λόγω της παρεμπόδισης εξάσκησης των ε, εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να ε, φέρουν εις πέρα στα καθήκοντά τους, δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ε, το δίκαιο δεν καθορίζει το πώς πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους οι τρίτες, τα τρίτα μέρη με τη ε, δύναμη κατοχή. Αλλά μπορεί κανεί να αντλήσει συμπεράσματα από τι σχετικέ συνθήκε και συμβάσει. Το πλέον σημαντικό είναι ότι η διαδικασία του συντονισμού πρέπει να είναι εύλογη, αποτελεσματική, να μην ε, επιτρέπει διακριτική μεταχείριση, αλλά είναι ζωτική σημασία σε αυτό ο μηχανισμό συντονισμού να διέπεται από την καλή πίστη, ώστε να μπορεί να ωφελήσει η ανθρωπιστική βοήθεια αυτούς που ακριβώς τη χρειάζονται περισσότερο. Προκειμένου να αντιπροσωπευτούν τα σημερινά προβλήματα, είναι σαφέ ότι οι μηχανισμοί συντονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια που χρησιμοποιούν, ε, ε, ε, που παρεμποδίζουν οι Ισραηλινέ αρχέ, δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια που προανέφερα. Αντιθέτω, διαπιστώνουμε διαρκώ ότι υπάρχουν παραδείγματα και περιπτώσει όπου οι Ισραηλινοί ε, ήρθαν σε αντιπαράθεση με τα κριτήρια αυτά, με τι δράσει του. Μια άλλη στατικική που παρατρύναμε να αναπτυχθεί ως έναν μηχανισμό για να εμποδίσουμε την καταστροφή των ε, κατοικιών κυρίως στον τομέα ΣΥ ήταν ο χροταξικός σχεδιασμός των Ισραηλινών να ακολουθήσει κάποια όπως ονομάστηκαν ε, βασικά σχέδια ή έστω μερικά σχέδια εντό εισαγωγικών. Αυτοί είναι μηχανισμοί στους οποίους ε, οι δυνάμεις κατοχής των Ισραηλινών Ε, σχέδια τα οποία είναι στρατηγικές που χρηματοδότησαν ως βασικοί δωρητές η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φορείς της. Αρχικά τα σχέδια αυτά έδιναν την εντύπωση ότι παρέχουν κάποια προστασία στις κοινότητες Παλαιστινίων με την ε, προστασία των κατοικιών τους από τους ε, στρατιώτες, από τις δυνάμεις κατοχής. Όμως στην ε, πραγματικότητα, λόγω των διαδικασιών στις οποίες ανατρέχουν οι Ισραηλινές αρχές για την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, οξύνεται ο κίνδυνος κατεδάφισης, καταστροφής των συγκροτημάτων κατοικιών εκτός των ορίων που αναφέρουν τα ειδικά σχέδια. Επίσης η διαδικασία χαρτογράφησης των σύνορων των ορίων αφήνει πολλές κοινότητες εκτός των ορίων. Δηλαδή εγκρίνονται αυτά τα προγράμματα εις βάρος άλλων και ολόκληρα τμήματα του πληθυσμού καταλήγουν να είναι ε, παράνομα. Οι υποδομές, οι κατοικίες, το τείχος, οι κοινότητες αυτές εξαναγκάζονται να διαπραγματευτούν με τις ελληνές δυνάμεις μέσω τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για να συνδέσουν λόγω χάρη το αποθηκευτικό τους δίκτυο, το υδροδοτικό του σύστημα με αυτό των ε, εντό εισαγωγικών νόμιμων ε, επικοιών. Και επειδή αυτά τα βασικά σχέδια έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό και υλοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν ορισμένα μόνον συγκροτήματα κατοικιών και αυτά προστατεύουν. Οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή δημόσια κτίρια αποκλείονται, όπως τα σχολεία. Δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και δεν επεκτείνονται αναλόγως. Επίσης, προκαλούν συνέπειες και ως προς το εξής. Η δυτική όχθη κατακαιρματίζεται. Τα εδάφη της δυτικής όχθης κατακαιρματίζεται. Δεν υπάρχει εδαφική συνοχή ή συνέχεια μεταξύ των όμοιων πληθυσμών. Έτσι, αυτό που θα έπρεπε να είναι μια στρατηγική απόφαση για να διαφυλαχθούν κάποια μέρη του πληθυσμού από τις δυνάμεις κατοχής, είναι ένα νομοφανές εργαλείο που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινές αρχές για να προκαλέσουν περισσότερους εκτοπισμούς. Για αυτούς τους λόγους υπάρχει ανάγκη για μια πραγματική επαναξιολόγηση της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και το κατά πόσον μπορεί να συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές στο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτές οι ε, δραστηριότητες, οι ενέργειε δεν πρέπει να ολοκληρώνονται διότι αντιφάσκουν πλήρως με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Οι κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συμμόρφωση με τα κριτήρια και τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου όπως επικαιροποιήθηκε το 2009 είναι ένα καλό σημείο φετηρία. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη όλα αυτά να λάβουν και επιχειρησιακή διάσταση. Πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο αναφοράς που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να δρουν εντός του γενικότερου πλαισίου της ΕΕ κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους βάσει τη Σύμβαση της Γενέβης και ως προς τις ευθύνες τους ενώπιον των τρίτων κρατών. Επίσης, δημιουργήσαμε μια σειρά από, αποθετικούς στόχους ε, που θα εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς, οι ευρωπαϊκές δράσεις συμμορφώνονται με τις διεθνείς αρχέ του ανθρωπιστικού δικαίου. Γι' αυτό ε, συστήνουμε την έναρξη έρευνα και ανάκριση, καθώ και την εξέταση του κατά πόσον ε, το χωροταξικό σχεδιασμό συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ώστε να βεβαιωθούμε ότι ανθρωπιστικό διεθνέ δίκαιο, όπω ε, προβλέπεται στο σχεδιασμό τη πολιτική στην υλοποίησή του συνεχίζει να συμφωνεί με τι αρχέ του διεθνού δικαίου. Το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το Ισραήλ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δύναμη κατοχής και πρέπει να ε, απαιτήσει την άμεση πάυση οποιασδήποτε παράνομης κατεδάφισης. Θα πρέπει ως στρατιωτική αρχή να αναλάβει το Ισραήλ τις βασικές υποχρεώσεις του και να προσφέρει, την, ε, να καλύπτει τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Θα πρέπει η προσφορά βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχεται με προσοχή. Και πρέπει να ξεκαθαριστεί στην ε, κυβέρνηση των Ισραηλινών ότι οι περιοχές που κατέχει και οι κοινότητες που βρίσκονται υπό την κατοχή τους πρέπει να προστατεύονται πρέπει να απαιτηθούν αποζημιώσεις και εγγυήσει για το τι θα γίνει με τις δημεύσεις ε, και την κατάσχεση ε, ε, υποδομών ή τις κατεδαφίσεις υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτής της σημαντικότητας της μελέτης. Τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Μπέρμαν έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση αυτή. Την κοίταξα, έτσι, συνοπτικά, την έκθεση αυτή από την ε, διακονία και βλέπω ότι έχουμε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι περίπλοκα θέματα, ασχολούμαστε με αυτά εδώ και χρόνια. Πήγαμε στην Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη, στη Λεωρίδα τη Γάζα, και κάθε φορά βλέπουμε την ε, δύναμη κατοχή να μην σέβεται τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις της. Κάθε φορά βλέπουμε ότι ο Παλαιστινιακός λαός στραγγαλίζεται και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά. Βλέπουμε την απελπισία, ε, ιδιαίτερα στα μάτια των νέων, που μεταναστεύουν για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Βλέπουμε αγρότες που δεν μπορούν να φτάσουν στην, ε, στη γη τους, να την καλλιεργήσουν. Βλέπουμε οικισμούς να καταστρέφονται, άλλους οικισμούς από την άλλη να μεγαλώνουν και ε, η βιωσιμότητα του Παλαιστινιακού κράτους είναι τουλάχιστον κατά με πολύ αμφίβολη. Και ο χάρτης αυτός ε, της Παλαιστίνης μου φαίνεται σαν παιδί με, με μαγουλάδες. Δεν βοηθάει, με ηλαρά. Τι να κάνουμε λοιπόν, να προσπαθήσουμε να υπάρξουν δύο κράτη ή να εγκαταλείψουμε όλη αυτή την ιδέα. Διότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν νομίζω να εγκαταλείψουν οι Ισραηλοί τους οικισμούς τους τόσο εύκολα και δεν νομίζω επίσης να μπορέσει να υπάρξει ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος που να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του πληθυσμού του στο μέλλον. Και για, σε αυτή την περίπτωση η λύση του ενός κράτους που θα εγγυάται ίσα δικαιώματα για όλους ίσως ήταν καλύτερη. Είναι φυσικά κάτι ουτοπικό την παρούσα στιγμή, αλλά εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Τεκεζέρη, το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τους δύο μιλητές για την παρουσίαση αυτής της μελέτης που πράγματι είναι μια επιπλέον μελέτη που αποδεικνύει πόσε είναι οι παραβιάσεις του ανθρωπιστικού, του διεθνούς μάλλον δικαίου στην πράξη. Επίσης <clears throat> δείχνει ότι η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μην προβλέψει οικονομικές συνέπειες για αυτές τις παραβιάσεις ε, του ανθρωπιστικού διεθνούς δικαίου, να μην ασκήσει δηλαδή πίεση στο Ισραήλ για να μην συμβαίνουν πλέον όλα αυτά. Πώς? Τι πρέπει να γίνει τώρα. Έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις, πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν και ευθύ εξ αρχής όλοι είναι αρκετά επιφυλακτικοί για αυτές τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω καμία άποψη, διότι όσο βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αξίζει τον κόπο, ούτε καν να φανταστούμε τι θα μπορούσε να συμβεί. Και μάλιστα τι θα μπορούσε να συμβεί αν αποτύχουν. Μοιάζει να είναι αυτή η τελευταία ευκαιρία να έχουμε μια λύση για δύο κράτη. Με δύο κράτη. Όταν όμως ακούω τι λένε οι ειδικοί περί δικαίου γύρω μου, μία ενδεχόμενη συνέπεια από την αποτυχία, την ενδεχόμενη αποτυχία αυτών των ε, διαπραγματεύσεων θα ήταν η διεθνής κοινότητα να αρνηθεί από εδώ και στο εξής, να ε, ενισχύει βοηθώντας την Παλαιστίνη. Δηλαδή να αναλάβει αυτά που αναλογούσαν στο Ισραήλ ως δύναμη κατοχής. Το έχω ακούσει πολύ να το λένε αυτό γύρω μου. Δεν μπορούμε να συναντήσουμε, να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, με την Συρία, με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να χάνουμε. Εφόσον δεν υπάρχουν και στην πράξη χειροπιαστές βελτιώσεις. Μισό δις ευρώ σχεδόν ετησίω ε, που στην Παλαιστίνη. Θα ήταν δραματικό αυτό, κάτι τέτοιο για του Παλαιστινίους και κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλούσε συνέπειε σοβαρότατε επιτόπου και με περιπτώσεις βίας. Παραδόξως όμως είναι μία από τις ενδεχόμενες συνέπειες. Η δεύτερη, και εδώ θέλω να λάβω αφορμή από όσα είπε και ο συνάδελφος, για τα κούμενα λέγοντα και εδώ, εάν αποτύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, Πράγματι, λένε όλοι, ε, επιστρέφουμε στην ε, λύση και στην ιδέα του ενός κράτους. Πολλοί μου λένε ναι, αλλά ένα κράτος με το ίδιο δίκαιο, τους ίδιους νόμους και για τα δύο μέρη, Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, δηλαδή να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα σε ένα κράτος με δύο πληθυσμούς. Αλλά όταν ε, πηγαίνω εκεί και επισκέπτομαι τη χώρα, είναι ακόμη πιο τοπικό αυτό από το να απαιτούμε δύο κράτη. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια αραβική μειονότητα ε, εντό των συνόρων του 67, ε, τα σύνορα του Ισραήλ δηλαδή, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Το να ζητούμε λοιπόν τέτοια δικαιώματα για όλου δεν είναι ακόμη πιο τοπικό από το να ζητούμε δύο κράτη. Δεν υπάρχει και καμιά φοβερή διαφορά τελικά, ούτε η λύση του ενός κράτους φαίνεται να μας ε, επιτρέπει να φανταστούμε κάποια πρόοδο. Γιατί τουλάχιστον η άλλη λύση μας επιτρέπει μια άμεση υλοποίηση. Για σας που τα μελετήσατε όλα αυτά, πώς φαντάζεστε ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο που είναι τόσο γνωστό. Με περισσότερη τόλμη, περισσότερες πιέσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσπαθήσουμε να φοβήσουμε χρησιμοποιώντας τα εμπορικά του που έχουμε στα χέρια μας ή να αφήσουμε τους Παλαιστινίους χωρίς βοήθεια και να έχουμε μια τρίτη Ιντιφάντα, έναν ιεροπόλεμο με τέτοιε τραγικέ συνέπειε, όπω αυτή που θυμόμαστε από την προηγούμενη, τη δεύτερη, που ήταν πολύ βίαιη. Η τρίτη θα είναι ακόμη σοβαρότατη. Πώ βλέπετε τα πράγματα. Ωραίε είναι οι διαπιστώσει, αλλά πέραν αυτού, εντάξει θα μου πείτε εσεί οι πολιτικοί πρέπει να αποφασίσετε, όμω ε, αυτά έχουμε στα ενωπιών μα να αντιμετωπίσουμε. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Κυρία ευχαριστώ πολύ. Είμαι από την Αντιπροσωπεία για την Παλαιστίνη. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και για την έκθεση. Έχω μιλήσει με κάποιους από εσάς και σας γνωρίζω. Και Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε τις πληρωμές. Ε, ακούγεται συνέχεια αυτή η ιστορία. Ορισμένες φορές ε, χρησιμοποιείται και το σλόγγαν «We're payers, not players». Αλλά το θέμα είναι ότι η Γάζα είναι υποκατοχή, υποπολιορκία και αυτό δεν φαίνεται να ενοχλεί το Ισραήλ, ούτε καν τον υπόλοιπο κόσμο. Υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και νομίζω ότι αυτό δεν συνάδει με τις αρχές μας ακόμα και αν συνάδει με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Ίσως λοιπόν δεν θα μπορούσε να είναι αυτή η λύση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Σε ένα ψήφισμα της αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη είχαμε κάνει έκκληση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων, διότι αυτοί τι κάνουν, κατεδαφίζουν και κατασκευάζουν καινούρια. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να πούμε αρκεί θέλουμε τα χρήματά μας πίσω. Και επομένω, εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους. Είναι χρήματα των φορολογουμένων αυτά και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το πει και η Επιτροπή Ανάπτυξης. Και όταν υπήρχε και μια αποστολή μια αντιπροσωπεία ε, το 2012 τη επιτροπή ανάπτυξη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κατασπατάληση τη αναπτυξιακή βοήθεια. Χρειάζεται καταπηγόντω ανθρωπιστική βοήθεια και όχι αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό, διότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανάπτυξη δεδομένων των συνθήκων. Ίσως λοιπόν η Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πού χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Αν παραβιάζονται οι κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά και να ζητηθούν ευθύνες από το Ισραήλ. Διότι δεν χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά, τα δικά μας χρήματα με σωστό τρόπο. Και θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι εμείς ε, λύσει πλέον των δύο κρατών. Απλώς υπάρχει μια κατάσταση ενός κράτους αυτή τη στιγμή και κατά την άποψή μου δεν αποτελεί λύση το ένα κράτος. Ε, θα οδηγήσει στον όλυθρο. Δεν είναι λύση, δεν ξέρω τι θα γίνει σε μερικές δεκαετίες, αλλά τη σήμερα ημέρα δεν είναι λύση. Το να έχουμε δύο-τρεις κατοίκους στον τομέα Α και να προσπαθούμε λίγο να τους... Ε, βολέψουμε όλους από τη μια και από την άλλη. Ε, αυτό είναι το σχέδιο του Σαρών άλλωστε. Και πραγματικά δεν θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε και αυτή την πρόταση που κάνουν ότι αυτό θα είναι το τέλος του Ισραήλ. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια λύση και για το Ισραήλ. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης να πιέσει κι άλλο για τις συμφωνίες ε, σύνδεσης. Διότι η παραβίαση του άρθρου 2, αν δεν κάνω λάθος, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και ταυτόχρονα θα πρέπει να περιμένουμε και το Ισραήλ τι θα κάνει, διότι εάν αποτύχουν και πάλι διαπραγματεύσεις, τότε είναι βέβαιο ότι η Παλαιστίνη θα προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη και θα ζητήσει καθεστώς μέλους και όλα τα υπόλοιπα και ούτω καθεξής στα Ηνωμένα Έθνη και θα προσφύγουν και στο δικαστήριο be helpful in that situation if they... Και ίσως εδώ θα ήταν χρήσιμο να πάνε το Ισραήλ στα δικαστήρια. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα νομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να μην χρησιμοποιήσουμε στρατηγικές ε, μποϊκοτάζ, αυτά θα τα αποφασίσει η κοινωνία των πολιτών. Εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα ένομα μέσα. Και χρειαζόμαστε και την καλή δουλειά που κάνετε εσείς. Και μία επιπλέον ερώτηση. Τι αντίδραση είχαμε από πλευράς Ισραήλ στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα λάβω εγώ τώρα το λόγο. Συμμετείχα και εγώ στην αντιπροσωπεία που μετέβη στην Παλαιστίνη και στη Γάζα και ήταν εντυπωσιακό το να διαπιστώσουμε ιδίως η την ε, απομόνηση την οποία έχει επιβάλει ουσιαστικά το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό λαό. Και το θέμα είναι πώς γίνεται να χρησιμοποιούν παρονόμως ε, τα κονδύλια για το χωροταξικό σχεδιασμό για να καταπιέζουν του Παλαιστινιακό λαό. Και αυτό το οποίο είναι σαφές ε, για μένα είναι ότι αυτό το οποίο ε, τα φέραμε να κάνουμε εδώ και δεκαετίες, δηλαδή να δίνουμε ανθρωπιστική, κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία είναι το ίμιση της βοήθειας που δίνεται στη Γάζα και στην Παλαιστίνη και είμαι της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, είναι παράλογο αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή ε, καταστρέφονται ακόμα και δικέ μας εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα λοιπόν να σα ζητήσω κατά πόσον θεωρείτε ότι τα μέτρα μποϊκοτάζ ε, θα αρχίσουν να έχουν συνέπειες στα κατεχόμενα εδάφη. Έχω δει κάποιους υπολογισμού που έκανε ακόμα και το ίδιο το Λικούντ, το οποίο ε, υπολόγισε τι θα στήχιζε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση εφήρμοζε ε, τα μέτρα της ε, στην πράξη και νομίζω ότι προβλέπεται ένα κονδύλιο της τάξης των 4 δις ετησίων και υπάρχει και η δήλωση η οποία λέει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία αυτή τη φορά και, τα, οι Ηνωμένε Πολιτείες θα προβλέψουν μέτρα μποϊκοτάζ. Ε, θεωρείτε ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν και θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή ε, έχουν γίνει δυσθεώρητα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Λάουρα Φαλαβολίτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Διακονία για την παρουσίασή της και ευχαριστούμε και για την έκθεση. Έχουμε μια πολύ ακριβή ανάλυση του χωροταξικού σχεδιασμού και της διαδικασίας αδειοδότησης του Ισραήλ. Ξέρουμε ότι υπήρξε ανάπτυξη σε χωροταξικό επίπεδο και Αυτά φυσικά είναι απαραίτητα και για την ανάπτυξη του Παλαιστινιακού κράτους. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ο στόχος της ε, συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Παλαιστίνη είναι να δημιουργηθεί κατάλληλη βάση για να υπάρξει το μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος. Μέχρι λοιπόν να ε, πάψει να θεωρείται βιώσιμη η λύση των δύο κρατών, αυτό είναι ο στόχος της συνεργασίας μας. Η σημασία του τομέα C για την ανάπτυξη του παρελιστινιακού κράτου στο μέλο είναι ζωτική και αυτό φυσικά επιβεβαιώνεται και από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και από την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας στην οποία αναφερθήκατε και φυσικά αυτό είναι και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη του τομέα C. Πέρσι, της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ, Ξέρουμε ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη του τομέα C έχει επικριθεί, διότι κατά κάποιο τρόπο υπονοεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το παράνομο καθεστώς αδειών το οποίο εφαρμόζει το Ισραήλ στο τομέα C. Αλλά Ξέρουμε ότι δεν είναι η απόλυτη λύση και δεν είναι η τέλεια προσέγγιση, αλλά θεωρήσαμε ότι είναι η καλύτερη λύση ε, προς το παρόν και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να έχουμε μια προσέγγιση χωρίς συγκρούσεις με τις Ισραηλινές αρχές ε, για τα κατεχόμενα εδάφη. Καταρχάς, ε, Αυτό προήρθε ως απάντηση στην Παλαιστινιακή Αρχή και επειδή η αναπτυξιακή πολιτική ε, ήταν συγκεκριμένη για την Παλαιστίνη, θέλαμε αυτό που ήθελε και η Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή, να μην υπάρξει άμεση αντιπαράθεση με τις Ισραηλινές αρχές ε, στα κατεχόμενα εδάφη, αλλά επίσης ένας από τους λόγους είναι ότι ο στόχος αυτού του αναπτυξιακού προγράμματος στον τομέα C στον οποίο υπάρχουν προβλέψεις για βοήθεια και στήριξη της, της τοπικής κοινότητας ε, ε, για να μπορέσουν να αναπτύξουν ε, σχέδια τα οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ισραήλ για να μπορέσουν ε, να κατασκευάσουν κατοικίες. Υποτίθεται ότι ο στόχος λοιπόν είναι ο αυτοπροσδιορισμός, ...στο να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτά τα εδάφη και να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή τη γη. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι και συμφωνούμε ως προς το γεγονός ότι ε, το καθεστώς το οποίο εφαρμόζει το Ισραήλ είναι παράνομο. Ο στόχος λοιπόν είναι να βοηθήσουμε τα τοπικά συμβούλια Και αυτά τα σχέδια τα οποία υποβάλλονται στις ε, Ισραηλινές αρχές Εμείς από πλευράς μας δεν περιμένουμε να υπάρξει ρητή έγκριση. Συμφωνήθηκε από τα κράτη-μέλη και από άλλους διεθνείς φορούς, φορείς ε, και την κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιείται στην Παλαιστίνη να υπάρχει μια καταληκτική προθεσμία εντός της οποίας εάν το Ισραήλ δεν απορρίψει ρητό στα σχέδια αυτά, θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί. Επρόκειται λοιπόν για συμβιβασμό κατά κάποιο τρόπο. ώστε να μην δεχτούμε πλήρως αυτό το καθεστώς με τις άδειες που ήθελε να επιβάλλει το Ισραήλ στην περιοχή αυτή. Τώρα, ε, για κάποια σχέδια σε πιο ευαίσθητες περιοχές, αυτά δεν υποβάλλονται καν στις αρμόδιες αρχές στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν 90 σχέδια εν εξελίξη. Και για πολλά από αυτά η προθεσμία των 18 μηνών έχει ήδη εκπνεύσει Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει η κατασκευή εντός του έτους. Βεβαίως εδώ προβλέπεται και διαπραγμάτευση και αντιπαράθεση με την GOGAT και ε, λαμβάνεται υπόψη και το θέμα της κατεδάφισης, διότι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι υπόλογη στους πολίτες της ε, για την κατεδάφιση εγκαταστάσεων ή οικοδομών οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και ο λόγος για τον οποίο ή μάλλον διορθώνει ομιλήτρια θεωρήσαμε ότι αυτός είναι ένα από του τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα κτίρια δεν θα κατεδαφιστούν από τις Ισραηλινές αρχές. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Διακονία για την ανάλυση. Νομίζω όμως ότι τελικά η απόφαση για να προχωρήσουμε με την προσέγγιση αυτή των σχεδίων, αυτών των master plans, ήταν μια απόφαση η οποία προήλθε με σύμφωνη γνώμη αρκετών κρατών μελών και ε, από το γεγονός επίσης ότι η τοπική κοινωνία είπε ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του τοπικού πληθυσμού στον τομέα σας. Ευχαριστώ πολύ. Merci. la... Ευχαριστούμε. Τώρα να δώσω το λόγο στους δύο εμπειρογνωμονές μας, για δύο λεπτά ο καθένας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Πέντε λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορώ μέσα σε πέντε λεπτά. Ε, θα αρχίσω με μια ερώτηση που ετέθη δύο φορές για τα δύο κράτη και ποια είναι η απόψή μας. Εμείς ως κέντρο έρευνα διεθνούς δικαίου θα θέλαμε η πολιτική συζήτηση να επεκταθεί λίγο και να δούμε, ε, να δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Και να θυμίσω στην Επιτροπή αυτή ότι ε, οι δυνάμεις κατοχής έχουν κάποιες υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Τώρα, ό,τι και να υπάρχει μέσα στο ψήφισμα από πλευρά πολιτικών συμβιβασμών, υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα που έχει ο πληθυσμός, ο κατεχόμενος πληθυσμός και αυτά τα δικαιώματα δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς. Ούτε η ΠΕΛΕ, ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτά λοιπόν είναι τα δικαιώματα που έχει, είχε και πάντα θα έχει ε, αυτή η ομάδα του ε, πληθυσμού. Προστασία δηλαδή και οι εκτοπισμοί και οι καταδαφίσεις απαγορεύονται, διότι υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις που το επέτρεψαν αυτό. Τώρα, όσον αφορά την άσκηση πίεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν πράγματι υποχρεώσεις ως τρίτα κράτη. Τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη προστασίας και διασφάλισης της ε, προστασίας του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτές είναι βασικές υποχρεώσεις και δεν τίθεται θέμα συμβιβασμών εκεί. Είτε αν αυτό είναι Παλαιστίνη, είτε αν αυτό είναι Σουδάν, Νότιο Σουδάν, η κατάσταση είναι η ίδια. Όσον αφορά το Διεθνές Παιδικό Δικαστήριο τώρα, ως νομικός οργανισμός εμείς ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να κυρώσουν τι συνθήκε, το καθεστώ τους. Πιστεύουμε πως έχει να δώσει προστιθέμενη αξία στις ειρηνευτικές διαδικασίε και να αποτελέσει καλό παράδειγμα και καλό προηγούμενο. Τώρα, οι ερωτήσει ε, τη ε, κυρία Σέλλορ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, υπάρχουν ορισμένα master plan που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όποια και αν είναι αυτή η απέτηση στο master plan, εάν αφαιρεί κάποια δικαιώματα από τον κατεχόμενο πληθυσμό, δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί στη συνθήκη της Γενέβης, οι... τα αιτήματα αυτά δεν ισχύουν, δεν έχουν καμία ισχύ. Και το πρόβλημα με αυτά τα σχέδια, με αυτές τις κατασκευές, είναι ότι βασίζονται στην μείωση του αριθμού των κατεδαφίσεων που θα γίνουν. Και μετά υπάρχει και ένα κριτήριο 18 ε, μηνών που πρέπει να περάσουν μέχρι να εγκριθούν αυτά τα σχέδια και μετά οι κατασκευές αυτές θα εγκριθούν και θα πραγματοποιηθούν. Ωστόσο όμως οι κατεδαφίσεις θα γίνουν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και ποιες τώρα είναι οι ευθύνε των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς να διασφαλίζεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία γίνεται σεβαστή, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι υποχρεώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει και να απαιτεί εγγυήσει μη επανάληψης και έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημιώσει έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες πρακτικές. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό ω αφετηρία. Υπάρχει τώρα ένα άλλο πρόβλημα του πώς εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική. Το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα έχουν συζητήσει αυτές ε, τις ε, ε, πτυχές, αυτά τα ενδεχόμενα στα πλαίσια της διεθνούς πολιτικής. Όμως, αποτελέσματα δεν έχουμε δει ακόμα και αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Ισραηλινές αρχές έχουν καταφέρει να μεταδώσουν αυτή την ευθύνη προστασία στη διεθνή κοινότητα. Την ευθύνη προστασία των ε, κατεχόμενων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Διεθνές Εθνικό Δίκαιο είναι ένα ουδέτερο δίκαιο είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να ε, μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε τις ε, πολιτικές. Είναι μια φορμή για συζήτηση και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που ε, χρησιμοποιούμε για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ και σε άλλες περιπτώσεις διενέξεων. Είναι καλή ιδέα η διεξαγωγή μια έρευνα, μια ανάκριση έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώ γίνεται με τον χώρο ταξικό σχεδιασμό του Ισραήλ. Θα ήταν, πιστεύω, ένα καλό τρόπος για να δούμε τι ε, ενδεχόμενε ε, συνέπειε. Όσον αφορά τώρα το να ζητήσουμε πίσω τα χρήματα που έχουμε δώσει συνάδει αυτό με την ε, οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη επανάληψη και για κατάσχεση ανθρωπιστικής ε, βοήθειας από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Βοήθειας. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο ομιλητές που μας έδωσαν κάποιες διευκρινήσεις για την παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και να περάσουμε τώρα η κυρία Ντεκεζέρ θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι δεν απάντησε κανείς την ερώτησή σας τελικά. Εσείς ρωτήσατε και δικαίως τι γίνεται με την πίεση που εξασκείται μέσω του μποϊκοτάζ ε, για ε, μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά είναι μια κατάσταση διακρίσεων και apartheid. Δικαίως λέτε ότι σήμερα από πλευράς της κοινωνίας των πολιτών υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση η οποία θα έπρεπε να προκαλεί όνειδος τουλάχιστον σε εμά τους πολιτικούς που έχουν και άλλα μέσα για να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Και είναι αλήθεια ότι σήμερα είμαστε μάρτυρες στη Γερμανία, σε πιέσεις στις τράπεζες που διαστηριοποιούνται στα κατεχόμενα εδάφη, ε, για επενδύσεις που γίνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα εδάφη, υπάρχει μποϊκοτάζ ε, ε στους επικισμούς ε, και ε, σε προϊόντα τα οποία προέρχονται από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους επικισμούς και ε, αρχίζει λίγο να ανησυχεί η Ισραηλινή κυβέρνηση ότι αυτό το κίνημα το οποίο ξεκίνησε από κάποιους ε, ε, στρατευμένους για το θέμα στην κοινωνία των πολιτών τελικά άρχισε να επεκτείνεται και γίνεται ένα πραγματικό όπλο για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Εμείς ε, ποτέ δεν έχουμε εκφράσει την απόψή μας εδώ στην Επιτροπή, γι' αυτό ακριβώς και παίρνω το θάρρος να επαναλάβω την ερώτησή σας, διότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέραν της ήπιας δύναμης έχουμε και άλλα μέσα για να ασκήσουμε πιέσεις. Και τι γίνεται με τα μέσα τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν σεβαστέ οι συμφωνίε οι οποίε έχουν προσυπογράψει τουλάχιστον. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ω μέσα πίεση. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Χρηματοδότηση ανάπτυξης. Έχουμε ζητήσει και αυτή τη μελέτη, την οποία θα μας παρουσιάσει ο κύριος Γκρίφιθ. Τον Ιούλιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση με τίτλο «Πέραν του 2015, μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση για την εκρίζωση της ένδυας και, τη βιώσιμη ανάπτυξη». Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, διότι ε, Υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες ε, σε διεθνές πλαίσιο εν εξελίξη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα το πάνελ υψηλού επίπεδου των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη μετά το 2015 και την ομάδα εργασίας και πάλι των Ηνωμένων Εθνών για τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ανακοίνωσής της εξετάζει τις διάφορες χρηματοδοτικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι, τόσο τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς, τόσο τους διεθνείς όσο και τους εθνικούς, όπως για παράδειγμα την φορολογία, τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις, τις δωρεές ε, φιλανθρωπικού χαρακτήρα και θέλει να αυξήσει τη χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη και να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στους στόχους που έχουν αποφασιστεί ώστε να είναι αποτελεσματική και συνεπής η πολιτική μας. Η μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή, η μας ε, θέλει να δει τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλει να αξιολογήσει και το έργο των Ηνωμένων Εθνών ευρύτερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ζητήματος περιττό να σας πω κύριε Γκρίφιθ ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε ε, τα όσα έχετε να μας πείτε για τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης σας και στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι της ε, Επιτροπής του ΟΣΑ και να δώσω λοιπόν καταρχάς ε, το, ρόλο στον κύριο Γκρίφι, το λόγο στον κύριο Γκρίφιθ για 10 λεπτά για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έκθεσης. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που είχαμε όχι μόνο να παρουσιάσουμε τη μελέτη αλλά και να την ε, κάνουμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνεργασία με τους χρηματοοικονομικούς εμπειρογνώμονες και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ορισμένα από αυτά τα σημεία που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να κάνω τέσσερα διαφορετικά πράγματα τώρα. Καταρχάς να σας δώσω μια γενική συνοπτική εικόνα ε, των πηγών χρηματοδότησης για την ε, ανάπτυξη και να σας ε, τονίσω τους κύριους στόχους. Έπειτα να συζητήσουμε τον, τον ρόλο της δημόσιας και της ιδιωτικής χρηματοδότησης στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Τρίτο, να συζητήσουμε την εμόκληση της ιδιωτικής χρηματοδότησης και γιατί παρουσιάστηκαν προβλήματα εκεί και ποιες είναι οι διαφορετικές αναλλακτικές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, τον ε, μελλοντικό της ρόλο από το 2015 και έπειτα στην στήριξη της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Εμείς θεωρούμε πως αυτό θα ήταν ε, καλή, πως αυτό θα γινόταν με τον καλύτερο τρόπο εάν εστίαζε στην δημόσια χρηματοδότηση. Αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα βασικά θέματα που θα σας αναφέρω. Τώρα, αρχίζουμε για τα, με τα τέσσερα βασικά γεγονότα, τις τέσσερις παραδοχές. Καταρχάς, ότι οι εγχώροι πόροι πρωτοστατούν στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Οπότε χρειάζονται λοιπόν αυτές οι επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν το 1 τρίτο του ΑΕΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε ότι ε, οι κυβερνητικές ε, δαπάνες παραμένουν οι κύριες δαπάνες. Ωστόσο, έχουμε 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε χώρες οι οποίες δαπανούν 3 δολάρια την ημέρα για να παρέχουν στους πολίτες τους τα αναγκαία. Παρότι λοιπόν οι κυβερνητικές δαπάνες ε, πρωτοστατούν είναι πολύ χαμηλές. Δεύτερη παραδοχή είναι ότι οι ροές προς τα έξω κονδυλίων είναι πολύ υψηλότερες από τις ε, ροές προς τα μέσα αποπληρωμές δηλαδή δανείων, για παράδειγμα το 2011 ανέρχονταν στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ε, επίσης έξοδος ε, ξένων επενδύσεων 420 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά λοιπόν είναι και μέσα σε αυτά υπάρχουν κονδύλια τα οποία έχουν αποκτηθεί παράνομα. 620 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ υψηλά ποσά τα οποία δεν έχουν ε, σε καμία περίπτωση χρησιμοποιηθεί με παραγωγικό τρόπο. Ε, τρίτη παραδοχή είναι ότι πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή όταν κοιτάζουμε τις εξενές επενδύσεις. Υπάρχουν ε, μεγάλες εκροές κέρδους, περίπου 90% του συνόλου των επενδύσεων, των εισερχόμενων επενδύσεων. Όμως από αυτό το ποσό το 60% είναι κέρδη τα οποία έχουν επανεπενδυθεί. Το 60% λοιπόν εκατό του συνόλου είναι χρήματα τα οποία έχουν ε, κερδιθεί σε μια αναπτυσσόμενη χώρα και έχουν επανεπενδυθεί σε αυτή. Δεν είναι λοιπόν καθαρή ισροή κεφαλαίων. Εάν λοιπόν συνυπολογίσουμε όλα αυτά θα δούμε ότι η επενδυτική αξία δεν έχει να κάνει τόσο με τα χρήματα που έρχονται αλλά με την ποιότητα των επενδύσεων που γίνεται, με το ποιε βιομηχανίε στηρίζουν αυτέ οι επενδύσει κτλ η αξία δηλαδή των επενδύσεων. Και η τέταρτη βασική παραδοχή είναι ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελεί την κύρια πηγή εισρωής ε, χρήματος. Ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλές δαπάνες. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μέρος της παρουσίασής μου. Ήταν τα τέσσερα βασικά σημεία τα οποία ε, περιέχει μελέτη μας. Το δεύτερο μέρος της μελέτης αφορά το, την δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση και το ρόλο τους. Δηλαδή, ε, με, την, ε, με τον όρο ιδιωτική χρηματοδότηση ε, αναφερόμαστε στα, στην χρηματοδότηση για κέρδη. Κερδοφόρο χρηματοδότηση. Καταρχάς να πούμε ότι η δημόσια χρηματοδότηση έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Στηρίζει την τα δημόσια αγαθά, παρέχει χρηματοδότηση για αναγκαίες ε, υπηρεσίες, ιδιαίτερα για τις ε, πιο φτωχές και περιοθωριοποιημένες ομάδες και χρειάζεται αυτή η δημόσια χρηματοδότηση για πάρα πολλούς τομείς, άμεση βοήθεια για παράδειγμα. Και αυτή πρέπει να είναι πιο σταθερή και σίγουρη από ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ε, έχει έναν σταθεροποιητικό ρόλο όπου εφαρμόζεται και είναι η μόνη πηγή ε, πόρων που έχουμε που απευθύνεται και μπορεί να απευθυνθεί στους φτωχότερε πληθυσμιακέ ομάδε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν πρέπει να ξεχάσουμε το ρόλο αυτό. Επίση, η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι επίση ιδιαίτερα σημαντική, έχει όμω περιορισμού. Για παράδειγμα, οι ξένε επενδύσει έχουν πολύ μικρότερο ρόλο ε, παίζουν πολύ μικρότερο ρόλο στις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες και είναι πολύ δύσκολο να στοχεύσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ε, πιο φτωχές αυτές χώρες. Και φυσικά υπάρχουν περιορισμοί σε, στις χώρες όπου υπάρχει ισχυρότερη δημόσια χρηματοδότηση για αυτές τις ε, πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Η δημόσια λοιπόν χρηματοδότηση έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και η ιδιωτική χρηματοδότηση περιορισμούς. Το τρίτο μέρος τώρα της παρουσίασής μου έχει να κάνει με την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε στην ιδιωτική χρηματοδότηση και υπήρξε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφερόταν σαφέστατα σε αυτά τα ε, θέματα και επίσης η ατζέντα για την ανάπτυξη προωθεί αυτούς τους στόχους, τη χρήση δηλαδή πιε, ε, ε, της άσκησης πίεσης στην ιδιωτική χρηματοδότηση για να βοηθήσουμε την δημόσια. Και εδώ ε, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα δεν είχαμε σαφή στοιχεία, γι' αυτό λοιπόν ε, παρατηρείται μια δυσκολία ε, στο να φτάσει η ιδιωτική χρηματοδότηση της σε μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Και ε, το ζητούμενο είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να δώσουμε προστιθέμενη αξία και να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά σε δημόσιες επενδύσεις που θα έπρεπε έτσι κι να έχουν γίνει. Έχουμε διάφορους ε, μηχανισμούς που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει κάποιους δείκτες για τις ε, λιγότερο ε, αναπτυσσόμενες χώρες, ένα καθεστώς, ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο θα συνδέεται με την χρηματοδότηση και θα βοηθήσει τις χώρες αυτές να ελέγχουν καλύτερα τους φυσικούς τους πόρους. Έπειτα υπάρχουν μέτρα για αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι οι πόροι αυτοί προέρχονται από δανεισμό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό επιφέρει και επιπρόσθετο κίνδυνο ε, χρέους. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι κίνδυνοι και στη μελέτη μας συνδέονται με το γεγονός ότι μάλλον δεν είναι και ο πιο κατάλληλος τρόπος να στηριχθεί μια φτωχή χώρα μια φτωχή χώρα η οποία έχει μεγαλύτερη ανάγκη από δημόσιες επενδύσεις. Το τέταρτο ε, σημείο που θα ήθελα να θίξω ήταν να προτείνω δύο ακόμα διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος, ενδεχομένως ε, μία λύση προς το πρόβλημα του πώς θα στηρίξουμε καλύτερα τις ε, οι ιδιωτικέ επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Καταρχάς θα πρέπει να αυξήσουμε τις δημόσιες επενδύσεις. Χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις στα σχολεία, στο παιδευτικό σύστημα, στην ε, περίθαλψη, στην, ε, στις μεταφορές, στις αναγκαίες ε, υπηρεσίες που αφορούν όλον τον πληθυσμό. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν, ότι όταν μιλάμε για τις δημόσιες επενδύσεις, που θα μπορούν να ασκήσουν πίεση στις ιδιωτικές, ε, πως αυτό είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα σε τοπικό επίπεδο όπου υπάρχουν είτε υπερβολικά πολλές είτε υπερβολικά λίγες πιστώσεις είναι πάντα προβληματική περίπτωση. Αυτό το έχουμε δει και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτό που λέμε στην ουσία είναι ε, μια επιστροφή στην παράδοση, στους παραδοσιακούς ε, τρόπους επενδύσεων. Και επίσης πιστεύω ότι στη μελέτη μας ε, φαίνεται πως λαμβάνονται μεν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη, όμως πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που έχουν στις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι σημαντικές αυτές ε, αποφάσεις είναι οι πολιτικές για την φοροδιαφυγή, για, τη, για την υπεύθυνη οικονομική διαχείριση και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσει θετικά την κατάσταση. Για παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει ε, για την οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος με τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων σε μια εταιρεία, έτσι ώστε να αποτραπούν οι μεγάλες απώλειες και η φοροαποφυγή, ιδιαίτερα σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα μέτρα που ενδεχομένως έχουν πολύ μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις από οποιασδήποτε αλλαγές στην πολιτική. Αυτά ήθελα σε γενικές γραμμές να πω και συμπερασματικά θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι εξίσου σημαντικές, έχουν διαφορετικό ρόλο η κάθε μία και χρειάζονται πλέον συζητήσεις για τις αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε στις δημόσιες επενδύσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκρίφιθ. Όντως έχουμε την αίσθηση ότι το κατέχετε το θέμα και είσαστε σε θέση να μας τα μεταδώσετε και με τρόπο εύληπτο. Οπότε ευχαριστώ και για τον τρόπο που εκφραστήκατε. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπεν από την Επιτροπή ΝΤΑΚ του ΟΣΑ. Καλησπέρα σας και όχι καλημέρα. Μου ζητήθηκε να σας μιλήσω για τα έργα της ΝΤΑΚ για την μέτρηση και την εξέλιξη της ε, εξωτερικής βοήθειας ε, και τις προβλέψεις για το 2015, μεταξύ άλλων η αναπτυξιακή αυτή επιτροπή του ΟΣΑ βασίζεται στην, ε, στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια για τις τρίτες χώρες και εργάζεται βάσει των δεδομένων που προβλέπουν οι, οι υποχρώσεις αναπτυξιακής βοήθειας με το 0,7% ε, του ΑΕΧ των, ε, των αναπτυγμένων χωρών. Πολλές φορέ υπήρχαν επικριτικά σχόλια με δαπάνες ε, των αναπτυσσόμενων χωρών που ποτέ δεν κοινοποιήθηκαν στις ανεπτυγμένες χώρες ή σε σχέση με την υποτίμηση των δανείων που έχουν παραχωρηθεί ως αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιούμε βασίζεται στις ροές μετρητών, δηλαδή την εξεκταμιεύση. Θεωρείται ότι υπάρχουν αρκετά κίνητρα ώστε να αναπτυχθούν ε, αναπτυξιακοί φορείς και να χρησιμοποιούνται και μέσα της αγοράς για την ε, ε, υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία όπως αυτά που βασίζονται στα αξιόγραφα ή η λεγόμενη χρηματοδότηση μετζανίν όπως ονομάζεται αλλά αυτά δεν είναι μετρήσιμα από την πλευρά της αναπτυξιακής βοήθειας λόγω του διαφορετικού κέρδους που μπορεί να προκύπτουν από την πώληση των αξιογράφων και από, από τον ενεχόμενο κίνδυνο το στατιστικό σύστημα δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτά τα εργαλεία, ούτε το παθητικό και το ενεργητικό και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από τη σκοπιά της ε, ροής μετρητού όπως εμείς καταγράφουμε πλέον τα δεδομένα. Το, στη συνάντηση της DAC με τη συμμετοχή ε, υπουργών υπεύθυνων για την αναπτυξιακή βοήθεια από το 2012 από τότε έχει ανατεθεί σε μας εντολή για ένα νέο εργαλείο της επίσημης, ε, για τη μέτρηση της επίσημης βοήθειας που παράσχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμπεριληφθεί σήμερα στις στατιστικές για την αναπτυξική βοήθεια. Ως μέρος της εντολής αυτής μας ζητήθηκε να κοιτάξουμε τις δυνατότητες να ε, περιγράψουμε καλύτερα και τη σκοπιά του δωρητού ως προς αυτά και όχι μόνο την πλευρά του κέρδους ε, των δικαιούχων. Διότι οι δύο αυτές κοπιές δεν ταυτίζονται απαραίτητος. Το τρίτο στοιχείο της εντολής που έχουμε είναι να εξετάσουμε κατά πόσον η νέα μέτρηση τη ε, επίσημης βοήθειας για την ανάπτυξη απαιτεί ε, εξυγχρονισμό και της παλιότερης μεθόδου μέτρησης λόγω χάρη με αλλαγέ στον τρόπο που εκταμιεύονται ή καταγράφονται τα δάνεια στο σύστημά μας. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο ε, έργο μπροστά μας και στον ΩΣΑ αρχίσαμε να επεξεργαζόμαστε τα ζητήματα αυτά. Έχουμε κάνει αρκετέ αναλύσεις και τις έχουμε αποστείλει στα μέλη μας για να τις εξετάσουν. Επίσης, ρόλος μας είναι να υποβάλουμε προτάσεις για ενδεχόμενες αλλαγές για το τι θα γίνει μετά το 2005 με το στατιστικό πλαίσιο του, της με βάση τις φετινές ε, μας διαπιστώσεις για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σφαιρικοί στην προσέγγιση μας. Είχαμε συζητήσεις και με άλλους φορείς, όχι μόνο με τους συνηθισμένους, αυτούς που συμμετέχουν στις συναντήσεις της ΝΤΑΚ στο Παρίσι και γι' αυτό δεχτήκαμε πρόθυμα και αυτή την πρόσκληση να σας μιλήσουμε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο να σας πω όλη την ουσία της δουλειάς μας σε λίγα λεπτά, αλλά αφού διάβασα τα έγγραφα που μοιράστηκαν ως ε, μελέτη υποστήριξη για τη συζήτηση αυτή, νομίζω θα τονίσω μερικά μονοσημεία. Το γεγονός ότι το σύστημα επιβολή στατιστικών εκθέσεων, σαν αυτό που χρησιμοποιούμε στον ΩΣΑ, είναι ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών για τα σχέδια του δημοσίου τομέα, του κρατικού τομέα, είτε για τα μεικτά οικονομικά μέσα, είτε για το σύστημα εγγυήσεων ή εξωγράφων. Από την άλλη, εφόσον συμμετέχει ο δημόσιο τομέας σε αυτές τις επιχειρήσεις, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες για την χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα γνωρίζουμε όλοι και νομίζω οι συντάκτε τη έκθεση που παρουσιάστηκε προηγουμένω θα συμφωνούσαν μαζί μου, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, δεν είναι επαρκή, ότι υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την ε, δίκηση και τη διακυβέρνηση και μπορούμε να εξετάσουμε έτσι τι διάφορε ροέ προ τι αναπτυσσόμενε χώρε καθώ και τον αντίκτυπο που είχαν. Ξέρουμε αρκετά για τι ροέ ε, ανθρωπιστική βοήθεια, ε, αναδραστηριότητα και ανατομέα. Αλλά δεν ξέρουμε πολλά για τι υπόλοιπε ροέ συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ξένη βοήθειας. Των άμεσων ξενών επενδύσεων μάλλον. Είναι άκρω εμπιστευτικές οι πληροφορίες αυτές για την ώρα. Ένας από τους στόχους λοιπόν που έχουμε για τη δουλειά μας στον ΩΣΑ είναι να διευκολύνουμε τη συλλογή αυτών των πληροφοριών που μας είναι απαραίτητες. από άλλες πηγές επίσημες εκτός της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πιστεύουμε ότι το να δημιουργήσουμε ένα σύστημα για να εντοπίσουμε αυτές τις πληροφορίες θα βελτιώσει τη λειτουργία μας για γιατί όλοι οι κυβερνητικοί φορείς και οι κυβερνήσεις μας εξήγησαν ότι δεν μπορούν πραγματικά να αξιοποιήσουν εργαλεία όπως αυτό των εξεγράφων και των μετοχών η των εγγύσεων, διότι αυτά πολλές φορές δεν καταγράφονται ω αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται στον ΩΣΑ είναι ότι τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να είναι εύστοχα σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες και ότι θα πρέπει να τα προωθήσουμε, αλλά καταγράφοντας πάντοτε και τις εισρωές και τις εκροές Συζητούμε λοιπόν ακόμη στον ΩΣΑ εάν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ε, στο νέο εργαλείο μέτρηση τη συνολική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια προ τι αναπτυσσόμενε χώρε. Κάτι ανάλογο με το εργαλείο που χρησιμοποιείται σήμερα για την καταγραφή τη αναπτυξιακή βοήθεια. Νομίζουμε ότι τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να ήταν χρήσιμα στι χώρε μεσαίου εισοδήματο. Εάν χρησιμοποιούνταν ευρύτερα μάλιστα για να δούμε την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε και στα εισοδήματα των ε, χωρών με χαμηλά εισοδήματα. Είναι πολύ η τεχνική μα δουλειά στον τομέα αυτό εδώ και ένα εξάμεινο και οι πολιτικέ συζητήσει μόλι ξεκίνησαν. Γι' αυτό με χαρά θα θέλαμε να, ακούσουμε τις απόψεις των διαφόρων ενδιαφερομένων και τις ε, θέσεις τους, ε, καθώς και τις απόψεις του Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ να ακούσουμε τις απόψεις σας λοιπόν για τα θέματα αυτά στην άλλη συζήτηση. Αν έχετε ερωτήσεις προς εμάς για τα δουλειά που κάνουμε στον ΟΣΑΘΜΟ με αυτό, παρακαλώ να μας τις θέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στην ε, κυρία Σαλντάνα από την Κονκόρντ ε, για πέντε λεπτά. Προηγουμένως όμως να καλωσορίσω τους φίλους της κυρίας Λέβιν. Είναι πολύ σημαντική για μας το Κοινοβούλιο. Πρέπει να σας το πω, γιατί έχει συμβάλει τα μάλα στην ε, υλοποίηση μιας νέας πολιτικής βιώσιμης αλίας. Δεν Κυρία Σαλντάνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου τη Concord για το επίσημο χρηματοδοτικό εργαλείο τη ΤΑΕΚ θα επανέλθω στα θέματα που ανέφτυξε ο κύριος Γκρίφης. Νομίζω ότι πραγματικά του αξίζουν ευχαριστίες αυτών και τους υπόλοιπους συντάκτες της έκθεσης για την εκπόνηση της μελέτης αυτής. Μετά από τις τελευταίες παρατηρήσεις του κ. Γκρίφη θέλω και εγώ να πω τα εξή. Όπως είπε, δεν υπάρχει ένα μόνο σημείο τη χρηματοδότηση τη ανάπτυξη. που μπορούμε να θεωρήσουμε ως τέλεια λύση. Και αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν διεθνείς συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει κατά πόσο η κρατική βοήθεια μπορεί να ενισχύσει τις ιδιωτικές προσπάθειες. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη λύση. Μαζί με τις προσπάθειες που μόλις σας απαρίθμησε ο Τζέσι, έχουμε δει ε, ελλείψεις και πλημεληματά στις προσπάθειες τη οικονομική παρέμβαση στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίω με την πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για την ανάμειξη. Στην Επιτροπή Ανάπτυξη είδαμε ότι δεν υπάρχει ακόμη επαρκή λογοδοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τι προσπάθειε αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και υπάρχουν τέτοιε απαιτήσει. Περισσότερη διαφάνεια λοιπόν στον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα δημόσια κονδύλια ω συνοδευτικό των ιδιωτικών. Αφού το είδου λοιπόν η δημόσια λογοδοσία θα πρέπει να είναι μέρος του κοινωνικού συμφώνου που ισχύει και εφόσον διευρυνθεί ο ορισμό τη αναπτυξιακή βοήθεια για να συμπεριλάβει τα ανάμεικτα οικονομικά μέσα, τα μεικτά μάλλον οικονομικά μέσα, την ιδιωτική χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό όμω να δούμε και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση τη αναπτυξιακή ατζέντα, όπω σωστά ανέφερε ο Τζέσι. Ένα σημαντικό θέμα για μα είναι και η κινητοποίηση των εγχώριων κοντιλίων, ε, δηλαδή οι προσπάθειε που γίνονται σε ε, εγχώριο επίπεδο για να υπάρξουν από την ιδιωτική αγορά ή δημοσίω και να εξευρεθούν κονδύλια. Υπάρχουν ε, δυσκολίες από την πλευρά των ε, κρατικών αρχών, υπάρχουν περικοπές, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες από τους ιδιωτικούς φορείς να βρουν τους πόρου που χρειάζονται σε εθνικό ή διεθνέ επίπεδο. Όπω ανέφερε εδώ ο Τζέσι, υπάρχουν συγκεκριμένε ευθύνε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το επισημάναμε και πέρυσι. Αποκρινόμενοι στην έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη, Financing for Development, αυτό το έγγραφο δηλαδή. Πέραν αυτού, νομίζω είναι σαφές στις διεθνείς συνομιλίες ότι μια συγκεκριμένη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με τις δεσμεύσεις της προς την ανατεξιακή βοήθεια. Όπως είπε ο Τζέσι, τα δημόσια κονδύλια και η εθνική ή η διεθνής βοήθεια διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες που αναφέρονται και στην έκθεση της Concord από πέρυσι. Σας προσκαλώ μάλιστα να την ξεφυλίσετε αν το έχετε κάνει ήδη. Μαζί με την εξέταση του την αντιπτυξική βοήθεια είναι σημαντικό να σκεφτούμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, αρρωγή. Προβλέπεται συνάντηση στο Μεξικό όπου θα εξεταστεί το θέμα της διεθνούς συνεργασίας για τα θέματα αυτά. Εκεί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει εκ νέου τις ευθύνες της, για να δεν επιλώνει τις υποχρεώσεις της και τις δεσμεύσεις της. Πέραν όμως αυτών υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση, με τον έλεγχο, με την διευθέτηση. Όλα αυτά επηρεάζουν την ικανότητα των χωρών να απορροφήσουν δημοσιογητικά κονδύλια, ώστε να είναι παραγωγικές και να καταβάλουν τι μέγιστε δυνατέ προσπάθειε για την ανάπτυξη. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα προσοχή. Παρακαλώ, απευθύνω έκκληση στο Ευρωκοινοβούλιο στη συζήτηση των θεμάτων αυτών να τα δείτε σφαιρικά όλα αυτά. Μην επικεντρώνεστε σε μια ή την άλλη πτυχή, αλλά να δίνετε την ίδια προσοχή σε όλα τα σημεία. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στα μέλη τώρα. Ο κύριος Μπέρμαν έχει τίσει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με χαρά αυτές τις τρεις αναλύσεις για το μέλλον της ε, χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Υπάρχει κάτι το οποίο προβλημάτισε και ίσως θα μπορούσε να με διαφωτίσει ο Τζέσι. Μας είπες ότι η μόχλευση της δημόσιας χρηματοδότησης είναι αμφισβητήσιμη όταν συζητούμε ιδιωτικά προγράμματα. Και ανέφερες, για παράδειγμα, το 1 προς 31, το οποίο σημαίνει περίπου 97% της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο. Μήπως ε, είναι λίγο βιαστικό αυτό το συμπέρασμα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν βέβαια η Δήμων, απλώς πολιτικός είμαι, ε, η δημόσια χρηματοδότηση ανοίγει το δρόμο και διασκεδάζει φόβους ιδιωτικών επενδυτών ώστε να ε, χρηματοδοτήσουν προγράμματα. Και ακόμα και αν η μόχλευση είναι πολύ μεγάλη, και μειώνει κατά κάποιο τρόπο την επιρροή των δημοσίων φορείων είναι σημαντική διότι έτσι επιτρέπεται στα προγράμματα να ε, υλοποιηθούν. Είναι λίγο αμφισβητήσιμο το να δηλώνει κάποιος ευθαρσός ότι εάν είναι μεγάλη μόχλευση ε, καλό θα, ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν έχουμε κανέναν άλλον που να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ξέρω για παράδειγμα ότι στην Ανατολική Ευρώπη με 30 εκατομμύρια ευρώ ως ε, εγγύηση πίστοση ε, χρηματοδοτούνται προγράμματα αξίας ενός 2,2 δισεκατομμυρίων και κάθε φορά αυτό ε, το μικρό ποσό χρησιμοποιούνταν ως εγγύηση για πίστοση. Δεν συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Αντιλαμβάνομαι βέβαια αυτό που λέει η Concord ότι η ιδιοκτησία της αναπτυσσόμενης χώρας και ο δημοκρατικός έλεγχος του δανεισμού είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα από ό,τι κάνουμε σήμερα. Και η Concord ε, συμμορφώθηκε προς αυτό το, στη διάρκεια του τελευταίου σύντου και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό σοβαρά. Αναφερόμαστε σε αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, δεν θέλουμε να μην υπάρχει διαφάνεια, ίσα ίσα θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Θα μπορούσατε λίγο να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα της μόχλευσης και να μου εξηγήσετε πού κάνω λάθος. Διότι νομίζω ότι κάθε δημόσιο ευρώ πρέπει να χρησιμοποιείται με φιδό και αν με ένα ή δημόσιο ευρώ μπορέσουμε να έχουμε 30 ιδιωτικά ευρώ, πολύ ευχαρίστω. Αλλά πέστε μου που κάνω λάθο. Ευχαριστώ, κυρία Σαρτζεντίνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κάθε φορά που ακούω κάποιους που θέλουν να ξεκινήσουν ε, στη συζήτηση για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, φοβάμαι. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιληφθώ λοιπόν αυτή την παρουσίαση των εκπροσώπων του ΟΣΑ, διότι κάθε χρόνο, κάθε φορά που συναντούμε δημοσιονομικά ελλείμματα στον αναπτυξιακό προπολογισμό των κρατών μελών, έρχεται κάποιος Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ε, ε, αποφασίζει ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσει την αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε η αναπτυξιακή βοήθεια να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και τούντες άσυλο ε, πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη. Εάν λοιπόν σε καιρούς οικονομικής κρίσης όπου διαπιστώνουμε ότι η συνολική αναπτυξιακή δαπάνη όλων των κρατών μελών μειώνεται. Εγώ είμαι από τις κατοχώρες, είχαμε πολύ καλό ιστορικό το οποίο χάθηκε και τώρα είμαστε στο 0,6% ενώ είχαμε 0,8% πριν από τρία χρόνια. Και αυτό το οποίο χάνουμε ποτέ δεν το ξανακερδίζουμε σε μια τέτοια συζήτηση. Αναρωτιέμαι λοιπόν πού θα μας οδηγήσει αυτή η συζήτηση στον ΩΣΑ για τον ορισμό της αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, υπό την ε, προϋπόθεση ότι υπάρχουν ε, θεμητές επενδύσεις και θεμητό εμπόριο, θα μπορούσαμε όντως να μην έχουμε αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά επειδή εγώ είμαι πολύ παραδοσιακή και θα ήθελα να μην πειράξουμε καθόλου έναν ορισμό για την αναπτυξιακή βοήθεια σε μια συζήτηση ε, ασφάλειας αντί ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη και τούμπαλιν, αυτό όντως ισχύει, αλλά πραγματικά θα ήθελα να ξέρω τι θα γίνει και τι συνέπειες θα έχουμε, έχουμε ένα νέο ορισμό. Και μια δεύτερη παρατήρηση για τον πρώτο μιλητή. Εγώ είμαι η για την αναθεώρηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Ε, υποτίθεται ότι θα γινόταν ψηφοφορία την Πέμπτη, θα αναβληθεί γιατί ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, για, αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, αλλά πραγματικά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή πλειοψηφία από όλα τα φάσματα των πολιτικών ομάδων. Βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά από όλε τι πολιτικέ ομάδε φαίνεται ότι είναι όλοι υπέρ των δημοσίων μητρών για του τελικού χρήστε και τελικού ε, ε, ιδιοκτήτε, και το γεγονός ότι θα υπάρχει ένα δημόσιο μητρό για μα είναι πάρα πολύ καλά νέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Φιώνα Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή συζήτηση, διότι προέκυψε από μια συζήτηση που έγινε εδώ στην Επιτροπή μας μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το 2015 σε μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση για την εκρίζωση της ένδυας και την ανάπτυξη και ε, εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες εκείνη τη συζήτηση και εγώ και ο συνάδελφος Γκέρνσον ζητήσαμε κατά πόσον θα μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία, διότι στην αρχική συζήτηση ε, μας ζητήθηκε η παρουσίαση και ευχαριστούμε πάρα πολύ που κανονίσατε να γίνει αυτή η παρουσίαση. Υπάρχουν κάποια θέματα κλειδί και με εντυπωσίασαν στα όσα άκουσα από τον Τζέφι Γκρίφιθς. Ε, Είπατε ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση δρά διαφορετικά από τη δημόσια χρηματοδότηση και κάνει διαφορετικά πράγματα, επομένως η μία δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο της άλλης. Η ιδιωτική χρηματοδότηση έχει μια τάση να στοχεύει σε διαφορετικούς ανθρώπους, ανθρώπους ε, που βρίσκονται σε χώρες με υψηλότερα εισοδήματα και ε, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι φτωχότεροι λοιπόν στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε χώρες ίσως όπου το επίπεδο της δημόσιας χρηματοδότησης και δαπάνης δεν είναι πολύ ψηλό, μάλλον δεν βοηθούνται και πάρα πολύ από την ιδιωτική χρηματοδότηση και αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση από πλευρά σας. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο μου τράβηξε την προσοχή είναι το γεγονός ότι ε, πολλοί από τους φραγμούς που ε, υπάρχουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε ιδιωτικές ξένες επενδύσεις είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς οι ευρωβουλευτές. Είπε η κυρία Σαρτζεντίνη για παράδειγμα ε, για την έκθεση που θα συζητήσουμε αργότερα η οποία είναι ε, σχετική με το αντικείμενο. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε για φοροδιαφυγή, για να υπάρχουν αναφορές, για να έχουμε καλύτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα λησμονούμε διότι εμέσω ε, βοηθούν και τη χρηματοδότηση και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο για την ανάγκη κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα δημόσια οικονομικά, διότι κάθε φορά που περιπλέκονται τα πράγματα ε, υπάρχει μία τάση να απομακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο και να μην υπάρχει έλεγχος από καμία πλευρά. Και αυτό φυσικά δεν ικανοποιεί σε καμία περίπτωση σε μία δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω για τη μελέτη αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική και πολύ επίκαιρη. Συζητούμε εδώ και καιρό ε, κάποιες μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν σε θέματα ανάπτυξης, στις σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα και στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Ε, σίγουρα είναι κατάλληλη στιγμή λοιπόν για αυτή τη συζήτηση, διότι Μας ενδιαφέρουν και οι στόχοι της ανάπτυξης μετά από τους 2015 και τι άλλο θα προκύψει από την όλη αυτή συζήτηση. Για να δώσω ένα πολύ απλό και σύντομο ορισμό, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κατατέξουμε σε τρία επίπεδα. Έχουμε καταρχάς τη φιλανθρωπία, τους ε, πολυεκατομμυριούχους, είχαμε και κάποιους από αυτούς που ήρθαν εδώ και μας μίλησαν για τα σχέδιά τους, ε, τις δωρεές τους, ε, τις εκκλήσεις που κάνουν και σε άλλους πολυεκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους. Και έχουμε και διάφορες εκθέσεις για την ανισότητα που επικρατεί ανά τον κόσμο, το, πάνω, το γεγονός ότι πάνω από το 50% του ακαθαριστών χάριου προϊόντος ε, ε παγκοσμίω ε, και τι γίνεται με αυτά τα ποσοστά. Το ιδιωτικό κεφάλαιο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να ε, έχουμε συνεργασία και υπάρχει και το εξή το οποίο υποστηρίζουμε εμείς πάντα από πλευρά σοσιαλιστών, η διαφάνεια. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να βρίσκεται στη βάση οποιασδήποτε συζήτηση. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον άξονα τη φιλανθρωπία που είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να λάβει και τι κατάλληλε διαστάσει. Και μετά βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Τι θα γίνει με την εισρωή όλου αυτού του ιδιωτικού κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πολύ μακρά πορεία Πρέπει να διανύσουμε όλη αυτή την απόσταση και να δούμε πώς θα συνεργαστούν όλα αυτά μαζί. Πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα επιχειρήσεις θα αρχίσουν βαθμιδών, να δίνουν λίγο-λίγο κεφάλαιο, να υπάρχει... Ε, κοινωνική, εταιρική ευθύνη, αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπαγρυπνούμε ευθύ εξ αρχή. Και επίση υπάρχει και αυτό το οποίο συζητούμε εμεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα του blending. Και εδώ μας απασχολούν τρία θέματα τα οποία είναι ουσιώδη. Και θα τα ήθελα να θέσω και ως ερώτηση κάποια από αυτά. Καταρχάς ο έλεγχος των αποφάσεων. Ποιος θα λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις. Δεύτερον, κάτι το οποίο μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Ίσως θα καταφέρουμε μεγάλο τμήμα αυτών των χρημάτων να διατεθεί για μεγάλες υποδομές. Δεν ξέρουμε βέβαια ποιος αποφασίζει και πώς και χωρίς την κατάλληλη διαφάνεια πώς θα τα βρούμε αυτά. Και τρίτον, αυτό το blending και αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο και η ανάμειξη των δύο κεφαλών θα μας δώσει ε, κάποια ποσά τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να τα διαθέσουμε για άλλους στόχους και για άλλες προτε... προτεραιότητες στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Δηλαδή, να υπάρχει ένα ιδιωτικό, ε, ατομικό επίπεδο πολύ σημαντικό, ένα δημόσιο και παγκόσμιο επίπεδο το οποίο ε, έχει πολλή δουλειά, τι θα γίνει με την ε, διαφάνεια η οποία προχωράει πάρα πολύ αργά, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει αυτό το blending, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αναμίξουμε όλα αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Ευχαριστούμε. Και τώρα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σόρ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, ομιλητές, όλους τους συμμετέχοντες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Όπως ήδη αναφέρθηκε από, και από τους προηγούμενους ολιμητές, αυτή η εφαρμογή των συστήσεων για τη χρηματοδότηση είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο των εργασιών μας εδώ στις Βρυξέλλες και όπως ε, είπα πριν ψήφισαμε μια ανακοίνωση ε, για το τι θα γίνει μετά το 2015, για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρηματοδότησης ε, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Σχεδιάσαμε λοιπόν μια συνολική εικόνα του πώς θα μπορούσε να είναι αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σχέδιο από το 2015 και μετά και ποιες ε, αρχές θα ακολουθήσει. Είχε καλή αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους και τον ε, Δεκέμβρη υιοθετήθηκε ως συμπέρασμα του ε, Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν είναι η αρχή και η αφορμή για να αρχίσουμε τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Ξέρω πως ε, η Επιτροπή Ανάπτυξης δεν είχε την ευκαιρία να αναλύσει και να συζητήσει την ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής, ωστόσο πολλά μέλη από αυτήν εδώ την Επιτροπή είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την παρουσίασή μου στα πλαίσια της ε, Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Και θα ήθελα να κάνω κάποια έτσι, προκαταρκτικά σχόλια ε, για αυτή την μελέτη, γιατί δεν προλάβαμε να την κοιτάξουμε ενδελεχώς. Καταρχάς, να πω πως ε, καλωσορίζουμε αυτήν την ε, βάση για συζήτηση με αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Είναι δεδομένα που θα μας βοηθήσουν. Είναι καλή αφορμή λοιπόν για περαιτέρω εξέταση και είναι και, και όλα σε πολύ κοντά σε αυτά που κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασχολούνται με πολύ σημαντικά ζητήματα την χρήση των κονδυλίων και την ε, η διοχέτευσή τους. Η ιδιωτική χρηματοδότηση ανέρχεται στο 1 έβδομο της συνολικής χρηματοδότησης που πηγαίνει ε, σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα λοιπόν από τα κυριότερα μηνύματα της ανακοίνωσης είναι ότι πρέπει να δούμε ως πακέτο τη χρηματοδότηση και να δούμε την διαφορετική προσέγγιση ανά χώρα της βοήθειας αυτής. Η ανακοίνωση της Επιτροπής έχει καλύψει τα περισσότερα ζητήματα στα οποία αναφέρεται και η μελέτη. Όμως, σε αντίθεση με αυτή, δεν έχουμε κάνει προτάσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάσαμε, όμως, στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και περιεκτικής προσέγγισης μετά από συζήτηση με τους κοινωνικούς μας εταίρους. Τώρα, επί της ουσίας, συμφωνούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ε, ρόλο και τη σύνδεση ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση και στην ε, ανακοίνωσή μα αναφέρεται κιόλα η μεγάλη διαφορά ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση. Προχωράμε όμως και πέρα από αυτό, εξηγούμε τα κυριότερα εργαλεία που έχουμε για να δώσουμε κίνητρα για επενδύσεις και με μεγάλη χαρά βλέπω ότι η μελέτη αυτή συμφωνεί με πολλές από τις προτάσεις μας παρότι έχει ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση. Μας προβληματίζει όμως το ότι η μελέτη θεωρεί ένα πράγμα της δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Για παράδειγμα τα κυβερνητικά έσοδα δεν μπορούν να ε, αναλυθούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις και τα έσοδα από ιδιωτικές επενδύσεις. Διότι οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να αποφασίζουν για το πού θα δοθούν ευκαιρίες για ιδιωτικές επενδύσεις. Οι κυβερνήσεις όμως δεν μπορούν να επηρεάσουν το πού θα δοθεί πού θα δοθούν αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ε, ιδιωτικές επενδύσεις από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό. Οι επενδύσεις ε, σε γενικές γραμμές θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την, ε, την παροχή δημοσίων αγαθών και την αναπτυξιακή πολιτική. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, όσους ε, συνεισέφεραν στην μελέτη αυτή, γιατί είναι μια πολύ καλή αφορμή για περαιτέρω συζήτηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ερευνά τρόπους ε, με τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση για δημόσιους σκοπούς. Και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θίξατε και εσείς σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Τζέσι Γκρίφιθ. Τέσσερα λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Νομίζω λίγια από αυτά αφορούσαν άμεσα εμένα, αλλά είναι πολύ καλό να ακούω τη θέση του Κοινοβουλίου για την ε, οδηγία απαγόρευση τη ε, νομιμοποίηση παρανόμων προσόδων. Ελπίζω να εγκριθεί και από το Συμβούλιο. Συμφωνώ με όλου του ομιλητέ που υπογράμμισαν το ρόλο του Κοινοβουλίου σε συζητήσεις πολιτικού περιεχομένου που γίνονται παραλλήλως και μπορεί να έχουν ε, μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το θέμα της μόχλευσης λοιπόν ή της ανάμειξης ε, με ιδιωτικά κονδύλια και μέσα. Ο συνάδελφος από την Επιτροπή είπε ότι η έκθεσή μας συστήνει ότι πρέπει να συνδυαστούν τα δημόσια με τα ιδιωτικά κονδύλια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Λέμε πάντοτε ότι η δημιουργία κεφαλαίου, έτσι όπω την καταμετρούμε εμεί, δεν κάνει διάκριση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών κοντιλίων. Είναι δύσκολο να ξέρουμε ποιο μέρο τη εγχώρια επένδυση κάθε φορά είναι δημόσια ή ιδιωτική προέλευση. Αυτό είναι το μόνο χειροπιαστό στοιχείο. Ε, για μας αυτά έρχονται από κοινού ω προ τη μόχλευση. Θα ήθελα εδώ να πω τρία πράγματα. Πρώτον, ότι θεωρώ ότι είναι καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη οι δημόσιοι φορείς να σκεφτούν πώς μπορούν να κινητοποιήσουν, να επιδοτήσουν ή να βελτιώσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις σε κάποιες στις ε, διάφορες χώρες, αλλά πρώτα απ' όλα σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό οι διάφορες κυβερνήσεις να έχουν ισχυρές πολιτικές για το πού θα θέλουν να, να κατευθύνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις, με τι κριτήρια την ε, ε, προωθούν και τι ροές υπάρχουν, αν λόγου χάρη υπάρχουν καλύτερες ροές τη στιγμή που ξεσπά μια κρίση. Είναι στοιχεία που οι κυβερνητικοί φορείς πρέπει να τα δουν αυτά. Όμως οι συνομιλίες που προβλέπονται για το 2015, για το τι θα γίνει μετά το 2015, δεν λαμβάνει δεν, γίνεται, μάλλον, δεν γίνονται από τη σκοπιά του εθνικού ε, επίπεδου, της εθνικής διάστασης, αλλά από την πλευρά των πολυμερών, ε, των διεθνών οργανισμών ή της ευρωπαϊκής τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ή οι πολυμερείς θεσμοί δεν έχουν τον ίδιο σχεδιασμό με το τι, που να ανταποκρίνεται στο τι συμβαίνει στην πράξη. Η μικρή λοιπόν συμβολή του καθενός μπορεί να έχει οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη κίνηση και χρηματοδότηση, αλλά δεν είναι πάντοτε βέβαιο ούτε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Λόγου χάρη ο φορέας της ειδικής κυβέρνησης ετοίμασε μια έκθεση που υπολογίζει ότι 8 από 12 εταιρείε που επένδυσαν στην αναπτυξική βοήθεια θα το είχαν, δεν θα το είχαν κάνει χωρίς την ε, δημόσια μόχλευση. Και το 55% των επενδύσεων από ιδιωτικέ εταιρείε ω τώρα φαίνεται ότι θα είχε προχωρήσει χωρίς την κρατική στήριξη. Δεν ξέρουμε λοιπόν κάθε φορά ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν λέμε ότι θα υπάρξει μόχλευση με αυτόν τον τρόπο ή με την ε, ανάμειξη οικονομικών μέσων θα πετύχουμε καλύτερους στόχους. Δεν το ξέρουμε. Ούτε μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα γίνει ε, στην πράξη. Μόνο εκ των υστέρων μπορούμε να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα της δράσης μας. Νομίζω είναι σημαντικό πολιτικό ζήτημα αυτό για το Κοινοβούλιο και είναι σοβαρό να δούμε τι γίνεται με τα χαρτοφυλάκια των περισσότερων ευρωπαϊκών ε, φορέων αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Βεβαίω στηρίζουν τι επενδύσει από τι δικέ του χώρε ή τουλάχιστον τι χώρε του ΩΣΑ. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτή η στήριξη πηγαίνει όντω στην αναπτυξιακή βοήθεια ή αν υπάρχουν εθνικοί λόγοι να στηρίζει ο καθένα τι δικέ του εταιρείε που θέλει να επενδύουν. Είναι δύσκολο να τα σταθμίσει κανεί αυτά. Σε γενικέ γραμμέ πάντω νομίζω ότι πρέπει να αντιστρέψουμε την οπτική μα γωνία και να δούμε τι θέλουν οι αναπτυσσόμενε χώρε και εκεί να τι στηρίξουμε παρά να προποθέτουμε ότι έχουμε την απάντηση με του φοβερού μηχανισμού που προβλέπουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπέν για τον ΟΣΑ και την Επιτροπή ΝΤΑΚ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στην ερώτηση για την αναπτυξική βοήθεια και τις ενδεχόμενες αλλαγές στην καταμέτρησή της, τον υπολογισμό. Θα ήθελα να το δούμε από μια άλλη προοπτική το θέμα. Στον ΩΣΑ, αυτό που συζητήσαμε ξεκινήσαμε να συζητάμε, το ερώτημα που θέσαμε ήταν πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα κινητοποιήσουμε αρκετά κονδύλια για την ανάπτυξη μετά το 2015. Το γεγονό ότι επίση η αναπτυξιακή βοήθεια, όπω την ξέρουμε σήμερα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λύσει όλα τα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών στον κόσμο, ήταν κάτι που το επαναρχόταν διαρκώ στι συζητήσει μα εκεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εμπλέξουμε και τον ιδιωτικό τομέα του κοινού αναπτυξιακού μας στόχου. Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Και ω την καταμέτρηση, τον υπολογισμό, την παρακολούθηση του πώ εξελίσσονται τα προγράμματα του δημόσιου τομέα με τη μόχλευση του ιδιωτικού, είναι θέματα που μα απασχόλησαν ευθύ εξ αρχή. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά με την συνολική στήριξη, τη χρηματοδότηση που μπορεί να κινητοποιείται μέσω των επίσημων παρεμβάσεων, των κρατικών παρεμβάσεων. Ένα άλλο στοιχείο που δεν αναφέρθηκε ακόμη σήμερα. Είναι το, η διάσταση της ασφάλειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ειρήνευσης. Αυτά ακούστηκαν βέβαια, αλλά στον όσα διαρκώς αναφερόμαστε και στις διαδικασίες που ισχύουν μέσω του ΟΗΕ για μετά το 2015 για το σχετικό αναπτυξιακό πλαίσιο και τους αναπτυξιακούς στόχους για μετά το 2015. Ένα σύστημα που θα προσωμίζει σε αυτό του όσα θα βοηθούσε στην παρακολούθηση της χρηματοδότησης για τον διτό αυτό στόχο, εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία επί των στόχων. Αλλά σήμερα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε ακόμη. Διότι δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι που θα τεθούν μπορεί η ασφάλεια να είναι μια μεγαλύτερη προτεραιότητα τελικά. Αλλά ακόμη δεν μπορούμε να προβλέψουμε επιπλέον δαπάνες από την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα φανεί τι θα γίνει ε, εφόσον καταρτιστεί το σύνολο των στόχων που θα παρέχονται και θα καλύπτονται μέσω της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Και μια τρίτη παρατήρηση για την αναπτυξιακή βοήθεια και πάλι. Συζητήθηκε το κατά πόσο πρέπει να έχουμε αυστηρότερα μέτρα ε, και τρόπους υπολογισμού από ό,τι στο παρελθόν προσέξαμε από το τι ίσχυσε στο παρελθόν με την υποβολή εκθέσεων ότι υπήρχαν μέθοδοι καταμέτρησης που άφηναν μεγάλο περιθώριο ερμηνεών. Και υπήρχαν σοβαρές αποκλήσεις στον τρόπο που τα μέλη της ΔΑΚ κατέγραφαν τις ροές, τις δαπάνες τέλο πάντων, στα συστήματά μας. Η συζήτηση λοιπόν που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το τι μπορούμε να κάνουμε για να αποσαφηνίσουμε τις ε, κατατήρες γραμμές που έχουν δοθεί και η καταμέτρηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας να είναι αξιόπιστη και να πείθει και το κοινό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ολοκληρώσουμε τώρα με την κυρία Σαλντάνα για να ολοκληρώσουμε με τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι, διότι μας δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσουμε από πλευράς της Concord. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν ε, στη διάρκεια της συζήτησης. Καταρχάς για να ενισχύσω αυτό το οποίο σας είπα, το επιχείρημά μου δηλαδή ότι δεν υπάρχει χρυσή λύση στην ε, αναπτυξιακή ατζέντα. και όλη αυτή η διαδικασία για το πώς ε, θα είναι η συνεισφορά στην αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς θα προσμερτήσουμε, για παράδειγμα, την βοήθεια που γίνεται για τη μεταρρύθμιση των ε, διαφόρων κυβερνήσεων, που είναι προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να υπάρχουν ε, ένα κατάλληλο πλαίσιο χρηματοδότησης μετά το 2015 και τι γίνεται με τους κανόνες εμπορίου και επενδύσεων που επηρεάζονται πάρα πολύ από την ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Και αυτή είναι πολύ σημαντική πτυχή της χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ατζέντα και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τα επαναπροσδιορίσουμε ή να τα έχουμε όλα προσμετρήσιμα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μετρήσουμε ποσοτικά, αλλά είναι μια εξίσου σημαντική πτυχή της όλης συζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να την παραγνωρίσει και να μην δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν θα είναι στα πλαίσια της ε, ε, χρηματοδότησης και το αναπτυξιακό θεματολόγιο μετά το 2015. Τα είδαμε αυτά και στην ατζέντα του G20. Πόσο είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει και να προχωρήσει μια πολύ σημαντική πτυχή της ε, χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Το γεγονός δηλαδή ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να πρέπει να αντιμετωπίσουν τους ε, αθέμητους κανόνες που χρησιμοποιούνται στο νομισματικό σύστημα και τι γίνεται με την υποτίμηση και την υπερτίμηση ορισμένες φορές ε, λόγω συγκεκριμένων δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται διεθνώς ε, και διαφόρων διευθετήσεων στο νομισματικό σύστημα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά τη μόχλευση. Για να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Μία ακόμα σημαντική πτυχή, ε, η οποία αναφέρεται στην έκθεση, είναι το πώς θα μετρήσουμε επακριβώς πώς η δημόσια χρηματοδότηση και η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόχλευση για συγκεκριμένε επενδύσεις σε αναπτυσσέμενες χώρες που θα έχουν στη συνέχεια πραγματική ανάπτυξη. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μόχλευση αυτή τη στιγμή είναι προς ε, μεγάλα έργα υποδομών. Δεν υπάρχει βέβαια απαραίτητος καμία απόδειξη ότι αυτό ε, συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη και αυτή είναι μια πτυχή την οποία θα πρέπει επίσης να προσμετρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την σημαντική συνεισφορά σας ε, στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, Να περάσουμε τώρα στο σημείο 9 της της διάταξης. Καινοτομία στην Επιτροπή μας συζήτηση των τροπολογιών έκθεσης. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες οι οποίες υπευλήθησαν στην έκθεση της κυρίας Αργεντίνη για την πρόθεση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των εξορρεκτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στην κυρία Σαρτζεντίνη για να μας παρουσιάσει εντάχει τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι στο σχέδιο εκθεσής της και να υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία είναι αύριο. Ναι κύριε Πρόεδρε, όντως θα ψηφίσουμε το θέμα αυτό αύριο. Για να είναι ομαλή λοιπόν η ψηφοφορία, Συζήτησα με τους αδέλφου την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο προκειμένου να διευκρινίσουμε κάποιε από τις προτάσεις μου και να υπάρξει μια συνεννόηση και για τις δικές τους προτάσεις. 77 τροπολογίες είχαμε στην έκθεσή μου για την προώθηση της ανάπτυξη μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών στην εξορρυκτική βιομηχανία στι αναπτυσσόμενε χώρε. Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου προκαλεί τη μεγαλύτερη συζήτηση και νομίζω ε, πολύ εύγλωτα μου έθιξε και η Φιώνα Χολ, δεν υπάρχει ε, νομικά δεσμευτική εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τι εννοείται. Ναι, όντως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι οξύμερο το ο, όλο σχήμα νομική, δεσμευτική, εταιρική, κοινωνική ευθύνη αλλά νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές μορφές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην εξορεκτική βιομηχανία, αλλά επειδή όλα είναι επιθελοντικής βάσεως και ε, προκύπτουν από διαφορετικά θέματα, δεν υπάρχουν κάποιες κοινέ προδιαγραφές τις οποίες σέβονται όλοι. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε διεξόδους, ώστε να μπορέσω να συνεχίσω μια έκθεση η οποία παρακινεί να καταλήξουμε σε μία κοινή προδιαγραφή την οποία θα σέβεται όλος ο κλάδος και θα ήθελε αυτό να είναι και νομικά δεσμευτικό. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Με τη Φιώνα Χόλ λοιπόν, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια για τους φιλελευθέρους και το Φιλίπ Μπρουλάν, ο οποίο είναι σκιώδης για το ΕΛΚ, προσπάθησα να καταλήξω σε μια διατύπωση η οποία δεν θα είναι τόσο πράσινη και θα προσπαθήσει να συμπεριλάβει και όλες τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και όλα αυτά μέσω κάποιων συμβιβαστικών προτάσεων και προφορικών τροπολογιών. Αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω εδώ βέβαια είναι οι τροπολογίες για τα ορυκτά ε, τα οποία δημιουργούν ο Φίλιπ Κασμάρακ από το ΕΛΚ υπέβαλε τι σχετικέ τροπολογίε, ο κύριος Ντέβα από τους συντηρητικού και δημοκράτες. Δεν είναι παρόντες όμως, ελπίζω να είναι εδώ οι σύμβουλοι του, οι οποίοι μετά από τι συνεδρίσει θα μου εξηγήσουν τι ακριβώς είχαν κατά νου. Διότι εγώ τι βλέπω. Εγώ είχα ένα κείμενο Έχουμε λοιπόν την τροπολογία 66, 69, 71, 72, 74 και 75, οι οποίες τροπολογίες περιορίζουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και τις νομοθετικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για ε, ευρωπαϊκές ε, τέτοιες δυνατότητες. Αν δείτε όμως την πρόταση που έχουμε για τα ορεικτά αυτής της μορφής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιούν τα ίδια ε, ορυκτά που έχει και η αντίστοιχη νομοθεσία στις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι συγκεκριμένα μεταξύ των οποίων ο χρυσό. Υπάρχουν ελάχιστοι οι οποίοι κάνουν εξόριξη αυτών των ορυκτών. Έχουμε ένα στο Ιναυστρία, Αυστρία, έχουμε ένα για κασίτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πάρα πολύ περιορισμένα όλα αυτά. Και αν περιορίσουμε εμείς και τις προτάσεις μας ε, μόνο σε ανάντι νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει ότι κάθε παραγωγός οποιοδήποτε καταναλωτικού αγαθού που περιλαμβάνει ένα από αυτά τα τέσσερα ορυκτά τα οποία αποτελούν αντικείμενο σύγκρουσης, διαμάχης, δεν έχει να λογοδοτήσει πουθενά και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και να προστατέσουμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά θα ήθελα να μιλήσω και υπέρ των επιχειρήσεων. Θα ήταν ιδιαίτερα άβολο αν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έπρεπε εξορρυκτικής βιομηχανία να τηρήσουν συγκεκριμένη νομοθεσία όταν όλοι οι υπόλοιποι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποχρεωμένοι να τηρούν αυτέ τι κανόνε. Επομένω για μένα η ανάντη κατά η κατάντη νομοθεσία θα πρέπει να πάει από κοινού διότι δεν είναι δυνατόν να τι διαχωρίσουμε σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο ε, αφορά στο γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να μην υπάρχει αναφορά στην ε, αμερικανική σχετική νομοθεσία, το US.Frank, ε, θα ήθελα να του απαντήσω το εξή. Ναι, όντω δεν είναι πολύ καλή αυτή η νομοθεσία και οδηγεί και σε δυνατότητα εμπάργκο αλλά η ευρωπαϊκή νομοθεσία θέλει να βοηθήσει και τη βελτίωση της αμερικανικής νομοθεσίας. Και δεν είναι η ίδια νομοθεσία, αλλά θέλει να είναι συγκρίσιμη. Δεν θέλουμε να έρθει η Έριξον, η Philips, η Siemens, οι οποία θα είναι υποχρεωμένες να ε, ε, τηρήσουν δύο διαφορετικές νομοθεσίες, την αμερικανική και την ευρωπαϊκή. Αυτό δεν βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες και δεν βοηθά και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επομένως, επειδή η αμερικανική νομοθεσία ασχολείται με όλη την αλυσίδα διανομής, από το ορυχείο στον καταναλωτή. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι καλύτερη, να μπορέσει να βοηθήσει τα πράγματα και να ασχολείται με όλη την αλυσίδα διανομής από τον πρώτο εισαγωγέα, ο οποίος εισάγει πρώτη ύλη ή και το κατεργασμένο, επεξεργασμένο προϊόν το οποίο καταφτάνει από κάποιο παραγωγό στην Κίνα. Διότι εκεί παράγονται τα περισσότερα ε, αγαθά υψηλής τεχνολογίας. Η ερώτηση μου λοιπόν προς το ΕΛΚ και τους συντηρητικούς και δημοκράτες για αυτές τις τροπολογίες είναι είστε βέβαιοι όντως αυτό θέλετε ε, να γράψει η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για αυτά τα ορυκτά ε, και να κάνει, να περιορίσει τις δυνατότητες που έχουμε για τους ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό και να είναι υποχρεωμένοι μόνο αυτοί να τηρούν την νομοθεσία. Εμείς νομίζω ότι θα τους δυσκολέψουμε απλώς τη, δολή, τη ζωή. Δεν έχουμε τόσους πολλούς εδώ στην Ευρώπη, αλλά όλη η Νοτιοανατολική Ασία θα δράνε ενόχλητη, χωρίς καμία τιμωρία και υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες για ε, βιώσιμη εξόριξη χωρίς σε περιοχές εκτός συγκρούσεων που, σε όλο τον κόσμο. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Φιώνα Χολ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη και είχαμε λοιπόν επικοδομητικές και καρποφόρες συζητήσεις την περασμένη εβδομάδα. Καλωσορίζω αυτή την έκθεση, είναι φιλόδοξη, προωθεί ε, υπεύθυνε επαγγελματικέ πρακτικέ ιδιαίτερα στην εξορρυκτική βιομηχανία και είναι πάρα πολύ σημαντικό που εμεί ασχολούμαστε με αυτό πριν από την πρόταση τη Επιτροπή και ελπίζω η Επιτροπή να λάβει υπόψη τη τα αποτελέσματα τη εκθεσή μα εδώ. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με, τους, ε, με τον πλούτο των φυσικών πόρων και πιστεύω πως η χώρα που χαρακτηρίζεται περισσότερο από αυτό το πρόβλημα είναι η δημοκρατία του Κονγκό, η οποία είναι μια πάρα πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους χώρα, ωστόσο... Την τελευταία φορά που είδα τους εδείκτες ανάπτυξης ήταν στο, τελευταία θέση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η, η συγγήτρια ανέφερε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και νομίζω πως συνόψισε πολύ καλά τις δικές μου απόψεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω οι επιχειρήσεις να έχουν φυσικά υψηλά στάνταρτ, όμως η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι στην ουσία κάτι επιπρόσθετο που κάνουν οι επιχειρήσεις πέραν από τις νομικές τους υποχρεώσεις, από αυτά που πρέπει για το νόμο να κάνουν. Και οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω, να προβλέπεται από τον νόμο και αυτό πρέπει να το δούμε και αυτό το ονομάζουν εταιρική κοινωνική ευθύνη. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με αυτό αυτή τη στιγμή. Όταν μια εταιρεία ισχυρίζεται πως κάνει κάτι για το περιβάλλον, μπορεί να χρησιμοποιεί τελείως διαφορετικές μεθόδους και πρότυπα από μια άλλη. Γι' αυτό και στην, ε, στις τροπολογίες 14, 15 και 44 χρησιμοποιώ αυτά τα, αυτό τον όρο, τα ενιαία πρότυπα. Και ως μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επίσης, οι επιχειρήσεις ισχυρίζονται πως ε, κάνουν πάρα πολλά καλά πράγματα για το περιβάλλον. Και εδώ πέρα έρχεται αυτό το πράσινο ξέπλυμα. Ισχυρίζεσαι δηλαδή ότι κάνεις κάτι για το περιβάλλον, όμως ε, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό και πώς αυτό γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν έλεγχος. Τώρα κάτι άλλο που θα ήθελα να πω για την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ότι στην τροπολογία 45 θα προσπαθήσω να αλλάξω την αρχική διατύπωση. Προτείνω να υπάρχει αυτή η υποβολή εκθέσεων ως υποχρέωση σε, στις ε, συμβάσεις τους, οι συνθήκες τους και ζητώ αυτές οι συνθήκες να ε, ζητούν την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών εταιρική κοινωνικής ευθύνης από πλευράς των επιχειρήσεων. Τώρα κάτι άλλο σχετικά με την έκθεση της εισηγήτριας είναι οι φόροι εξαγωγών. δεν νομίζω πως θα έπρεπε να περιορίσουμε τους φόρους εξαγωγών και να λέμε ότι αυτές οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης πρέπει να απέχουν από την ε, επιβολή περαιτέρω φόρων. Πιστεύω ότι μόνο με το άνοιγμα της αγοράς θα καταφέρουμε να έχουμε καλές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, αλλά αυτό πρέπει να είναι αμφίδρομο. και το να ζητάμε από τις χώρες αυτές να μην επιβάλλουν φόρου φόρους εξαγωγών είναι κάτι που πρέπει να έχει και ανταπόδοση. Ιδιαίτερα όταν ε, τις περισσότερες φορές δεν μιλάμε και για μικρές αδύναμες χώρες, αλλά για ισχυρές χώρες όπως την Κίνα. Οι φόροι αυτοί εξαγωγών λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να αποτελέσουν ε, αντικείμενο άσκησης πίεσης και πιστεύω πως ε, θα ήταν ασφαλέστερο να μην επιμείνουμε στην, ε, στο σημείο αυτό για τους φόρους εξαγωγής. Ε, τώρα, συμφωνώ με την εισηγήτρια με το ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε χωρίς καμία συνέπεια τις εταιρείες που έχουν αυτή την πρακτική του downstreaming. ιδιαίτερα στον τομέα της ξυλίας. Πιστεύω πως ιδιαίτερα στον τομέα της ξυλίας υπάρχει ένα μεγάλο νομικό παραθυράκι που προκύπτει από αυτό το downstreaming. Και τέλος, να πω ότι δεν συμφωνώ με την τροπολογία 29 του ΕΛΚ για το ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ενημερώνονται για τα project που τρέχουν εκεί. Πιστεύω πως υπάρχει μεγάλη ενημέρωση και χρειάζεται συνένεση. Είναι ιδιαίτερη σημασία η συνένεση και η στήριξη των τοπικών αυτών κοινοτήτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υποφεληθούν οι μικρές αυτές κοινότητες από την ανάπτυξη. Έπειτα να πω ότι υπάρχουν κάποιες πολύ καλές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα μπορούσαμε να δούμε τι κάνουν ορισμένες εταιρείες και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Πάντως οι γενικές γραμμές ε, πιστεύω πως η έκθεση είναι πολύ δυνατή, θα έχουμε μια καλή ψηφοφορία αύριο και τη στηρίζω απόλυτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγο στον κύριο Κόρτε Λάστρα. Ε, ναι, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του σκιώδου συζητητή μα, του κυρίου Μάικολ Κάσμαν ο οποίος είχε πολύ στενή επαφή με την κυρία Σαριζεντίνη και με τους υπόλοιπους και όδους εισηγητές. Θα ήθελα εκ μέρους του λοιπόν να σας διαβάσω ότι συμφωνούμε με τη θέση της εισηγήτριας της κυρίας Σαριζεντίνη και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ούτε τις ε, τροπολογίες του ΕΛΚ ούτε τις τροπολογίες των φιλελευθέρων που θέλουν να άρουν τους δεσμευτικούς ε, όρους ε, και μάλιστα να εφαρμόζονται αυτά για όλα τα προϊόντα. Επομένως συμφωνούμε με την εισηγήτρια στη σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μικελάντζελο Μαργκερίτα για τρία λεπτά. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω απλώς το θέμα των ορυκτών των ε, συγκρούσεων στην έκθεση αυτή. Να ευχαριστήσω την κυρία Σαρχεντίνη για όλη τη τη δουλειά. όπω ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την υπατή εκπρόσωπο ετοιμάζει μια πρωτοβουλία σφαιρική για να ασχοληθεί με τα ορυκτά που βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων υψηλού κινδύνου. να σας πω τι είδους προβληματισμούς είχαμε αυτή μας απασχόλησε προκειμένου να αναπτύξουμε αυτή την πρόταση, διότι είναι πολλά τα αλληλένδετα ζητήματα, είναι πολλά από τα περίπλοκα σημεία, τα οποία πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του για να ασχοληθεί με τα μεταλλεύματα σε περιοχές ε, συγκρούσεων. Μιλήσαμε με προσώπους ε, της κοινωνίας των πολιτών, ε, των με κυβερνητικών οργανώσεων, του επιχειρηματικού κόσμου, μελέτη τεκτύπου που χρειάστηκε ένα χρόνο για να ετοιμαστεί, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείε και τι κόστο υπάρχει σε όλε αυτέ τι διαδικασίε. Πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε την πρωτοβουλία μα. Στο τέλο αυτή τη διαδικασία είχαμε επί τη ουσία έναν τριπλό στόχο. Ε, Τρει μάλλον στόχου που είναι καλό να του έχουν κατά νου ε, νομοθέτε στη δουλειά του. Πρώτον, προφανώ πρέπει η σχέση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων ε, και των, ε, της εμπορίας των ορυκτών πρέπει να διακοπεί. Αλλά και οι ευρωπαϊκές, οι αμερικανικές εταιρείες ή από άλλες χώρες θα πρέπει οι εταιρείες να μορφώνονται με τις κατευθυντήρες γραμμές που έχει δώσει στον ε, ΩΣΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλους. Είναι σημαντικό αυτό κατά την υλοποίηση των πρωτοβουλειών που έχουμε αγκρίνει. Τρίτος στόχο, τον ανέφερε και η κυρία Σαρχεντίνη και είναι ε, ύψη τη σημασία, πρέπει να περιορίσουμε τι τρευλώσει ε, στην αγορά. Στρεβλώσει που προκύπτουν από τι υπάρχουσε πρωτοβουλίε. Δεν λειτουργούμε σε ένα κενό, η Ντότφρανκ υπάρχει και η ζημιά έχει γίνει. Έχει γίνει λόγω της έλλειψης συμμόρφωσης. Ε, επειδή ακριβώς υπήρξε μια τάση διαφυγής από τις περιοχές ε, με προβλήματα, με συγκρούσεις. Τα συμπεράσματα λοιπόν αυτής της ε, συζήτησης και όλες αυτές τις μελέτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι πρέπει οι πρωτοβουλίες μας να βασιστούν, είναι μια μάλλον προσπάθεια από τις πλέον περίπλοκες που εμπλέκει όσο και πάρα πολλούς ενδιαφερομένους σε σχέση με άλλες και που μπορεί να χρειαστεί και μεγάλα σκέλη εξωτερική ανάθεση. Το τελικό μα λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την αλυσίδα παροχής στην πηγή της, διότι αυτό θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε διαφάνεια στις επιχειρήσεις. Ανέφερα τις πρωτοβουλίες του ΙΕ σχετικά. Δεν εννοώ όμως μόνο τους ε, ενδιάμεσους αλλά και τις εισαγωγές ορεικτών και μεταλλευμάτων. Όλες τις εισαγωγές μεταλλευμάτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε τα ανάλογα κίνητρα. Δεν είναι μόνο η νομοθεσία που δημιουργεί υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να δώσουμε τα ανάλογα κινήτρα στις επιχειρήσεις για να συμμορφώνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε ο μόνος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ ωραία. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Σαρχεντίνη και πάλι για να απαντήσει σε όλες αυτές τις φιλοφρονήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κόρτε Λάστρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ που έχετε τέτοια εμπιστοσύνη στην εκθεσή μου. Το εκτιμώ. Ευχαριστώ την Φιώνα Χόλ των Φιλελευθέρων που τόνισε ένα-δυο σημεία τα οποία τα συζητήσαμε έτσι κι αλλιώ όταν μιλούσαμε για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης θα ήθελα οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν εξαγωγικούς δασμούς αλλά όπως είπα και σε εσά και στο ΕΛΚ νομίζω ότι μια χωριστή ψηφοφορία θα ε, έλυνε το θέμα αυτό. για τα μεταλλεύματα, τα ορεκτά σε περιοχές συγκρούσεων. Νομίζω είμαστε πολύ δραστήριοι για το θέμα αυτό. Ε, πλέον, ε, είμαι από τους πλέον δραστήριους ε, στο Ευρωκοινοβούλιο και έχω συζητήσει με όλους όσοι ήταν ανοιχτοί για συζήτηση. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί η Γενική Διεύθυνση Εμπορία όταν λέει upstream. Τι εννοείται upstream. Εννοείται τις εισαγωγές οποιοδήποτε προϊόντος, αγαθού, οποιοδήποτε εξάρτημα εργαλείου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει τότε. Αλλά υπάρχουν οι απόψεις και θα παρακαλούσα το ΕΛΚ να το ξανασκεφτεί. Δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί στους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στους επενδυτές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να ξέρουν εάν επενδύουν σωστά. Δεν υπάρχει τρόπος να τους αποδείξουμε τι ακριβώς έχει κάνει ο υπεύθυνος τι έχουν κάνει οι υπεύθυνοι για την εξόριξη με τα Και παρακαλώ, ακούστε με, διότι δεν μπορώ να το παραβλέψω. Όταν μου λέτε ότι θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για το τι καταγράφουμε στις εκθέσεις, εάν πρόκειται για πρώτη ύλη, για επεξεργασμένο προϊόν, αυτό ήδη είναι μια πρώτη σκέψη, μια πρώτη λύση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περνούμε τώρα στο σημείο 10 της σημερινής διαταξής. Όχι να θυμίσω ότι η ψηφοφορία της έκθεσης αυτής θα γίνει αύριο στις 11 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Σας προσκαλώ να είστε εδώ. Περνάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων με τον Πολ Φρίξ του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Ο κύριος Φρίξ μας απέστειλε ένα κείμενο που αφορά την παρουσίασή του. Βλέπουμε εκεί τις απόψεις του όσα Και βλέπουμε κιόλα τι συμβαίνει με αυτό το κέντρο που κόστησε τόσα πολλά στου αλλά δεν έφερε ει πέρα στην αποστολή του. Σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε που καλέσατε τον ΩΣΑ να συμμετάσχει σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σε μια τόσο σημαντική στιγμή για το μέλλον τη αναπτυξιακή βοήθεια. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που καλέσατε το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και όχι τον ΩΣΑ στην ε, συζήτησή σας. Καταρχάς να σας πω ποιος είμαι. Στο Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων όπου εργάστηκα από το 90 ως το 95 μετά τις δυσκολίες μάλιστα που είχαμε το 2012 και ενώ είχα διευθυντικό ρόλο, αυτή τη στιγμή έχω απλώς ένα ε, προσωρινό συμβόλαιο, μια προσωρινή σύμβαση. Ε, η βασική μου εκπαίδευση είναι στην, στην οικονομία της ανάπτυξης και είχα εργαστεί και σε βελγικούς φορείς στο παρελθόν. Να σας παρουσιάσω το σχετικό πλαίσιο για τις συζητήσεις που προηγήθηκαν μας απασχολείται γίνεται με έναν κόσμο που αυτή τη στιγμή μεταβάλλεται και που οι άξονες διαρκώς ε, είναι, εξελίσσονται και είναι πολλαπλοί. Τις τελευταίες δεκαετίες λοιπόν βλέπουμε να μειώνονται οι πόροι κάποιων ανεπτυγμένων χωρών μεταξύ των οποίων οι ευρωπαϊκές καθώς και η αποτελεσματικότητά τους. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σαφές πλέον. Και οι αναπτυσσόμενες χώρες όμως έχουν ε, αλλάξει πάρα πολύ. Ορισμένες ακόμη πρόσφατα βρίσκονταν ε, στον ε, κατάλογο των χωρών με χρέη, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει σχεδόν ανταγωνιστές μας κάποιες από αυτές. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα κόσμο που αλλάζει και υπάρχει και ανταγωνισμός. Οπότε είναι φυσικό να θέτουμε το ερώτημα τι εργαλεία διαθέτουμε. Ποιο είναι το καταλληλότερο μέσο και τι ε, διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από τις εμπειρίες μας. Καταρχάς, να σας πω τι είναι το κέντρο επιχειρήσεων. Είναι ένας από τους δύο φορείς, μεικτούς φορείς που έχει δημιουργηθεί βάσει των συμβάσεων ε, του ΟΗΕ για την Κοτονού. δημιουργήθηκε το 1977 περίπου με τις ίδιες αρχές που δείπαν και το CTA, δηλαδή την ανάγκη εκφομηχανισμού των αναπτυσσόμενων κορών, την ανάγκη ανάπτυξης, ε, κάλυψης μάλλον των γεωργικών αναγκών, δηλαδή την επισητιστική ασφάλεια, αλλά και την ανάπτυξη του δυναμικού που αφορούσε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών. Πρόκειται για δύο παλιές πρωτοβουλίες που ουσιαστικά ήταν ε, αριλοσυμπληρούμενες στην αρχή. Ποια ήταν η αρχική αποστολή του κέντρου επιχειρήσεων. Θα τα δείτε και στις διαφάνειες. Πρόκειται κυρίως για τη βοήθεια προς τις μικρές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε δίκτυα που μπορούν να τις οδηγήσουν στον εκβιομηχανισμό τους, στην εκβιομηχάνησή τους μάλλον. Και ε, προκειμένου να υπάρξουν και μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίες. Αυτοί οι γενικοί άξονες φαίνεται να ήταν εύστοχοι, αλλά το τι έγινε εντωμεταξύ. μεταξύ. Στην εποχή, αυτή την πρώτη αυτή περίοδο που ήταν και η δική μου, ε, είχε 18 εκατομμύρια ευρώ στη διαθεσία του προπολογισμού το κέντρο επιχειρήσεων. Από αυτά τα 18 εκατομμύρια, περίπου τα μισά κατευθύνονταν προς τις επιχειρήσεις μας. Επιχειρήσεις και δράσεις σε 18 χώρες ΑΚΕ. Εάν διαιρέσουμε αυτόν τον επιχειρησιακό προπολογισμό για τον αριθμό των χωρών ΑΚΕ, δεν ήταν και πολλά τα κονδύλια που είχαμε. Οπότε ο αντίκτυπός μας ήταν λιγότερο αντίκτυπος χρηματικός παρά στον ρόλο της πρωτοπορίας που διαδραματίσαμε στην προώθηση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας και την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την ε, δημιουργία απασχόλησης καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας που πρέπει να περνά από τις επιχειρήσεις. Παίξαμε λοιπόν ένα ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό επί μία εικοσαετία χωρίς όμως να ε, ε, ανταποκρίνεται αυτό στα κονδύλια μας, τα οποία ήταν και περιορισμένα και ε, διασπαθισμένα. Και περιορισμένα μάλλον. που ήταν και περιορισμένα και διασκορπισμένα. Τώρα, ε, ο κεντρικός ρόλος των Βρυξελών ε, ήταν οι επικρίσεις μας για τον τρόπο που λειτουργούσαμε με τον περιορισμένο αντίκτυπο, τα λίγα αποτελέσματα που πετύχαμε να έχουμε. Χρειάστηκε λοιπόν να υπάρξει αποκέντρωση της λειτουργίας μας, κάτι που ξεκίνησε στη δεκαετία του προσπαθήσαμε να πάμε πιο κοντά στους ε, τελικούς ε, δικαιούχους, τις επιχειρήσεις δηλαδή. Γι' αυτό δημιουργήσαμε κάποιες ομάδες με επιχειρήσεις πιλότου στο Μπουρούντι, στον Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, στην ακτή του Ελεφαντοστού, με πολλές ε, μελέτες για μελλοντικές προβλέψεις. Μετά τη δεκαετία του 1990 όμως αυτή η αναπόφευκτη εξέλιξη για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα δεν συνεχίστηκε και μάλιστα επί σειρά ετών. Το κέντρο από την άλλη δεν ε, είχε διεύρυνση στην εντολή του στην αποστολή του. Θα έπρεπε όμως να φύγουμε από τον αυστηρό χώρο, τον, ε, από τον χώρο τον αυστηρό βιομηχανικό για να περάσουμε και σε άλλους τομείς. Το κέντρο λοιπόν επιχειρήσεων προσαρμόστηκε στις ανάγκες των ε, μικρομεσαίων ή τουλάχιστον αυτόν τον ε, στόχο είχε αρχικά. Δυστυχώς κάποια στιγμή τα πράγματα πήραν διαστάσεις ε, παράλογες καθώς η αποστολή μας διευρύνθηκε τόσο πολύ που οι σταδικές μας δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Θα έπρεπε δηλαδή να γίνουμε κάτι σαν ένας υπεροργανισμός για την ανάπτυξη, για τον ιδιωτικό τομέα και τους, ε, τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη. Θα ήταν ωραίο αν συνέβαινε αυτό, αλλά δεν συνέβη, διότι ακριβώ δεν αυξήθηκαν αναλόγω και τα κονδύλια του προπολογισμού μα. Με τέτοιε εντολέ λοιπόν, με τέτοια αποστολή, δεν γίνεται οι περικοπέ στον προπολογισμό να μην προκαλέσουν σοβαρού τριγμού και προβλήματα. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή, η, απο επικέντρωσή μας με κακές επιλογές, αφού δεν ενδιαφερθήκαμε για τις τοπικές πραγματικότητες, δημιουργώντας εγκαταστάσεις ώστε να είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις, με συνεργατικές ε, επιχειρήσεις, με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή τραπεζικά ιδρύματα που έπρεπε να στηρίζουν τους ε, δανειολήπτες. Πολλές φορές δεν έγιναν οι σωστές επιλογές στα σημεία τη της εγκατάστασής μας. Και από το 2007 τα πράγματα πήγαν χειρότερα. Υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στη διεύθυνση του οργανισμού μας. Σε 7 χρόνια είχαμε 7 διαφορετικούς διευθυντές. Εγώ είμαι ένας δυστυχής ε, απολολός ε, προσωρινός διευθυντής. Απολολός τρόπος του λέγει. Θα μπορούσα να είμαι. Το διαπιστώσαμε ότι το 40% του προσωπικού του κέντρου απολύθηκε με τρόπο όχι πάντοτε ιδιαίτερα κομψό, κάτι που προκάλεσε και πολλές ε, διαφορές, διαφορές που κόστισε πολύ να επιληθούν στο κέντρο. Κόστος που αναγκαστήκαμε να καταβάλουμε το 2013. Καταστροφικές λοιπόν μεταρρυθμίσεις το 2009 με περιορισμό της τεχνικής, ε, του τεχνικού δυναμικού που είχε αναπτύξει όσο το κέντρο. Ε, είχαμε στη διάθεσή μας συμβούλους πρώτης ε, τάξης, με, πολλά, με πολλές προοπτικές επιτυχίας. Εντάξει, θα επιταχύνω κύριε Πρόεδρε. Από το 2009 λοιπόν το κέντρο ουσιαστικά έχασε ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων τους. Γνώρισε κάτι σαν ακροτεριασμό. Αυτό λοιπόν προκάλεσε και περισσότερα προβλήματα στη λειτουργία του και τη διεύθυνση και το 2012 υπήρξαν δύο διευθυντές μέσα σε ένα χρόνο. Η κατάσταση ήταν πολύ, ε, ε, πολύ επικίνδυνη αυτή τη στιγμή το κέντρο επιχειρήσεων ε, δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αποκέντρωσής του, η οποία έγινε με βάση τις ε, τοπικές υπηρεσίες μας, αλλά το τοπικό επίπεδο δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς. Λείπουν ήδη οι πόροι για να προετοιμάσουμε το μέλλον μας και βρισκόμαστε σε μια περίοδο καθοριστική για, την επόμενη, για το επόμενο διάστημα. Οι περικοπές στον προπολογισμό το 2012, το 2013 και το 2014 έχουν φέρει το κέντρο σε μια κατάσταση αντικειμενικός ε, σταδιακής εξάλληψης, phasing out. Το γεγονός ότι το 2013 ο προπολογισμό μας έφτασε τα 1,3 για τις επιχειρήσεις μας, μόνο και μόνο για να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις μας που προβλέπονταν ούτως ή άλλως και με το 2014 μας βρίσκει με ακόμα περισσότερο μειωμένο προϋπολογισμό, όλα αυτά μας έχουν φέρει σε αδιέξοδο. Σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα, τον Ιούνιο του 2013, δημιουργήσαμε ένα blueprint, ένα κείμενο που καταγράφει την κατάσταση και τις απαρχές του προβλήματος και προσπαθήσαμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις, λογικές λύσεις, γιατί πάντοτε υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αναζητήσει κανείς λύσεις. Αλλά συνοπτικά, κυρία μου, και θα δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο έγγραφο που σας απεστάλλει, Καταρχάς πρέπει να καλυφθούν οι διαρθρωτικές μας ελλείψεις στη διακυβέρνηση. Το 90% των προβλημάτων του κέντρου οφείλονται σε ένα ελλειπές σύστημα διοίκησης και διακυβέρνησης. Ανα πάσα στιγμή αποφάσεις εκτός της σφαίρας αρμοδιοτήτων του κέντρου μπορούν να οδηγήσουν σε περικοπή του προπολογισμού. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε θα έπρεπε η Επιτροπή του ΦΕΝΤ... να παρεμβαίνει μόνο μία φορά με ένα οικονομικό πρωτόκολλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον προπολογισμό όπου συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι δανειστές μας δηλαδή και εκπρόσωποι των ε, ε, δικαιούχων, θα έπρεπε λοιπόν το σχέδιο προπολογισμού να εγκρίνεται από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και από ένα Συμβούλιο ε, σοφών θα έλεγα, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργούν σε γενική συνέλευση και να δίνουν την έγκρισή τους. Επιπλέον ε, θα έπρεπε να υπάρχει μια εντολή η οποία να αφορά είτε αμέσως το κέντρο είτε έναν διάδοχο οργανισμό. Εμείς προτείνουμε μια εντολή που να βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες. Τη διοργάνωση των τοπικών μας δυνατοτήτων προκειμένου να παρακολουθούμε στενά την δράση των επιχειρήσεων, την διευκόλυνση πρόσβασης στην χρηματοδότηση και στις αγορές. Επίσης, την διευκόλυνση της ανάπτυξης τοπικών υπηρεσιών. Θα πρέπει αυτό να γίνει για τα αμοιβαία συμφέροντά μα. Διότι η εταιρική σχέση χωρί αμοιβαία συμφέροντα είναι πλάνη. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε και να εμπλέξουμε και το δίκτυο των επιχειρήσεων καθώς και ειδικευμένε ε, οργανώσεις ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε ακριβώς την υλοποίηση της εταιρικής σχέσης και τις περαιτέρω επενδύσεις. Ε, το νέο αυτό προβλέπει ένα γενικό επιτελείο περιορισμένο. Περιορισμένο στις βασικές ανάγκες. Αξιολόγηση, έλεγχο, benchmarking, ε, δράσεις ε, πιλωτικές και αποτιμήσεις. Μια δομή αποκεντρωμένη, είτε ονομαστεί κέντρο επιχειρήσεων, είτε κάπως αλλιώς. Ένας οργανισμός δηλαδή που θα εξασφαλίσει τη διαδοχή του, είναι κάτι που θα πρέπει να αξιοποιήσει και νέες πηγές χρηματοδότησης. Να είναι αποτελεσματικό ο οργανισμό αυτός ως προς το κόστος και να δώσει πολλαπλά ωφέλη. Μια πραγματική αποκέντρωση, ποιοτική και ποσοτική, όπως έχει προταθεί, ώστε το κέντρο βαρύτητας του κέντρου να μετατοπιστεί προς την τοπική πραγματικότητα, προς τις χώρες δικαιούχου. αυτό είναι υψής της σημασίας. Ε, εν είδε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνοπτικά η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δύο επιλογές υπάρχουν και πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση. Είτε αναδιάρθρωση, εκβάθρων μεταρρύθμιση, όπως προτείνεται από το δικό μας αποτύπωμα, είτε ένα νέος, ένας νέος οργανισμός, ένα νέο μέσο. Αυτό που προτείνει λοιπόν το κέντρο είναι συμβατό και με τη δεύτερη λύση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όποια επιλογή και προκριθεί, υπάρχει το εξής μήνυμα που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Πριν πετάξουμε το μωρό μαζί με το νερό, θα έπρεπε να ε, μην ξεχνάμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Φρίξ που μας παρουσιάσετε την κατάσταση. Είναι περίπλοκα τα πράγματα για τον οργανισμό μας, για τον οργανισμό σας με, σοβαρά, ε, με δυσκολίες και με μεγάλο κόστος όμως. Λοιπόν, η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Φρίξ, σας παρακολούθησα. Δεν θα έλεγα αφοπλιστική η ειλικρινιά σας, αλλά δεν μας κρύψατε τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο θα ήθελα να καταλάβω. Η προστιθέμενη αξία της εμπειρίας σας εκ των έσω. Ακούσαμε για τις δυσκολίες, την κατάσταση που αντιμετωπίζετε και πρέπει να σας πω ότι όντως ήσασταν ιδιαίτερα ειλικρινείς ε, για το θέμα αυτό. Αλλά για να μπορέσετε να μας προσανατολίσετε ε, προς την ε, κατεύθυνση ότι πρόκειται για ένα κεφάλαιο στο οποίο πρέπει ε, να επενδύσουμε. Μας είπατε ότι έχετε κάποιες καλές ιδιότητες, αλλά δεν τις γνωρίζουμε. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο διαθέτεται, το οποίο είναι αναντικατάστατο σε σχέση με τους υπολείπους. Και ίσως να υπάρχει κάτι το οποίο εμείς ή τουλάχιστον εγώ δεν κατάλαβα εδώ. Δεύτερη ερώτηση. Η ερώτηση απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχει κάποιος. Τι έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά νου ε, για να σας αντικαταστήσει. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Ε, καταρχάς, ποια είναι τα βασικά σας καλά στοιχεία ποια είναι τα προσόντα σας και με τι θα μπορούσαν να σας αντικαταστήσουν. Αυτή η ερώτηση βέβαια απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πρόεδρος. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην Επιτροπή τώρα, η οποία θα μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Ο κύριος Πιέρα Μιλά, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε Φρίξ. Έχουμε μιλήσει διαμακρών ε, για αυτό το περιεχόμενο της πολιτικής στήριξης ε, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα κάνω τώρα εδώ ε, μια παρουσίαση του θεσμικού ιστορικού. Μια παρατήρηση να σας πω μόνο ότι η παλιά μέθοδος χάραξης πολιτικής ήταν κάθε φορά που υπήρχε ένα πρόβλημα να συστήνεται ένας νέος οργανισμός και να θεωρούμε ότι κάθε φορά που συστήσαμε τον νέο οργανισμό λύσαμε το πρόβλημά μας. Νομίζω ότι άλλαξαν οι καιροί. Ε, πρόκειται για μία μέθοδο η οποία ε, μάλλον δαπανηρή είναι τη σήμερον ημέρα και για τον προπολογισμό μας ε, και για όλους όσους τροφοδοτούν αυτό τον προπολογισμό. Και νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε στα συμπεράσματά του ο κύριος Φρίξ. Δηλαδή ότι ως προς την ουσία της πολιτικής στήριξης στον ιδιωτικό τομέα. Να υπενθυμίσω ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του θεματολογίου της αλλαγής, της ανάπτυξης. Προσπαθούμε να έχουμε τέτοιες πολιτικές. Ο κύριος Φρίξ στην ουσία στο τέλος μας είπε ότι πρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες στις επιχειρήσεις στις μικρές, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις μεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να τους παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες θα διευκολύνουν όχι μόνο την προσφορά, δηλαδή όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά και στήριξη στις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο μας ανέφερε είναι ότι χρειάζεται ένα δίκτυο επιχειρήσεων, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Φρίξ από αυτού, και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μας είπε, απαιτείται αποκέντρωση, συμφωνούμε απόλυτα επ' αυτού, και θεωρούμε ότι υπάρχουν και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ένα μακρύ κατάλογο για στήριξη στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα ήθελα τώρα να μακρηγορήσω, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά ναι, εμείς αυτή τη στιγμή ε, συνεργαζόμαστε με τη Γραμματεία των ε, χωρών ΑΚΕ, ε, την αρμόδια υπηρεσία εδώ στις Βρυξέλλες των χωρών ΑΚΕ, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει τις προτεραιότητες, ώστε να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για τις προτεραιότητες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη στήριξη στον ιδιωτικό τομέα. Ένα τέταρτο, πολύ σύντομα, η δημιουργία επιχειρηματικού ευνοϊκού περιβάλλοντος, δηλαδή να υπάρχει μια στήριξη ε, προς τις κυβερνήσεις μάλλον για την δημιουργία νομοθεσίας η οποία θα λαμβάνει υπόψη ε, και το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να απολευθερώσουμε κάποιες πρωτοβουλίες αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει και κατάλληλη νομοθεσία για τη διαφθορά και τη δικαιοσύνη. Να υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον λοιπόν και για τις επιχειρήσεις και για τις επενδύσεις ενα δεύτερο άξονα ε, να προτείνουμε υπηρεσίε. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριο Φρίξ, αλλά όντω χρειαζόμαστε υπηρεσίε και όσο πιο αδύναμη είναι μια επιχείρηση, όσο πιο μικρή είναι μια επιχείρηση, τόσο περισσότερε υπηρεσίε χρειάζεται σε επίπεδο ε, πολύ μικρών παροχών. Και η πρόσβαση στην, ε, στις μικροπιστώσεις, στη μικρή δανεδότηση. Θέλουμε να προτείνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ως μια ενιαία δέσμη μέτρων από πλευράς χωρών και θέλουμε να ασχοληθούμε με τις μικροπιστώσεις και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση λίγο πιο διαφοροποιημένα μακροπρόθεσμα. Αυτό το έγγραφο ετοιμάζουμε με τους συναδέλφους μας των χωρών και θα υπάρξει ένα κεφάλαιο το οποίο θα είναι ειδικά αφιερωμένο στις μικροπιστέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των γυναικών και στην απασχόληση των νέων. Ε, πρόκειται για συγκεκριμένο αίτημα το οποίο απευθύνουμε στους εταίρους μας από πλευρά ΣΑΚΕ και θα είναι η δεύτερη προτεραιότητα στην ε, ε μετουσίωση αυτής της πολιτικής. Ένας επόμενος άξονας είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάθε φορά όμως ε, δεν μας ενδιαφέρει απλώς και μόνο η προσφορά της χρηματοδότησης αλλά και η ζήτηση, δηλαδή να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να παρουσιάσουν προγράμματα τα οποία θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ε, επενδυτών. μια άλλη πτυχή είναι πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά και τι εργαλειοθήκη θα πρέπει να αναπτύξουμε προκειμένου να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Ε, θεωρήσαμε ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον μαζί με τις χώρες ΑΚΕ να ε, υπάρχει ένας μόνιμος διάλογος για τη στήριξη στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρούμε ότι αυτό το είναι το στοιχείο που λείπει, ο πολιτικός διάλογος για τη στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα μας επιτρέψει να καθορίσουμε μαζί με τους εταίρους μας και το περιεχόμενο των δράσεων που θα υλοποιήσουμε. Να τις ε, συνοδεύσουμε όλες αυτές οι δράσεις στο Δινεκές και να δημιουργήσουμε και μια κατάλληλη πλατφόρμα διαλόγου μαζί με τους συνομιλητές μας. Δηλαδή να μην ε, συζητούμε μόνο με τους εταίρους μας ε, από πλευράς χωρών και θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και η κοινωνία των πολιτών, η οποία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ρόλο, κυρίως στον τομέα των μικροπιστώσεων, αλλά και σε επίπεδο ε, ε, της συνδρομής στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ένα επόμενο στοιχείο αυτής της εργαλειοθήκης είναι να υπάρξει ε, ένας διάβλος ε, επικοινωνίας με τον ιδιωτικό τομέα για να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Η διευκόλυνση των επενδύσεων με την όλη συζήτηση που έγινε μόλις προηγουμένων κυρία Πρόεδρε είναι ε, δημόσιες επενδύσεις. Σε αυτές αναφερόμαστε. Θέλουμε στα πλαίσια αυτής της διευκόλυνσης των επενδύσεων ε, θέλουμε να κινητοποιήσουμε όχι μόνο ιδιωτικά κεμβάλα, ε, αλλά να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και ε, τις ε, δανειοδοτήσεις και τις επιδοτήσεις ακόμα και να έρχονται από το δημόσιο τομέα. Τρίτος άξονας δράσης, το να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις συμπράξεις με μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και αντίστοιχη σύμπραξη με την κοινωνία των πολιτών, στην οποία αναφέρθηκα, διότι ε, συμμετέχουν και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Τέταρτον, σε αυτή την εργαλειοθήκη, να δημιουργήσουμε ένα μέσο για τις υπηρεσίες τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Φρίξ. Δηλαδή να υπάρχουν ενδιάμεση ε, μεταξύ ε, των επενδυτών και των επιχειρήσεων, να δημιουργηθεί το κατάλληλο δίκτυο και όλα όσα ε, συνεπάγεται. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι η ανάλυση που έκανε ο κύριος Φρίξ με όλη αυτή την ειλικρίνεια όπως επισημάνετε κι εσείς ε, κύριε Ντεκεζέρ αλλά ίσως χωρίς όλες τις λεπτομέρειες που θα έπρεπε να αναφέρουμε για τη χρηματοδοτική πτυχή, ε, την περίπτωση της Όλαφ, ε, τι γίνεται με κάποια, κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να διαγραφούν. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε λοιπόν ότι το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να επιτύχει τους στόχους τους οποίους ε, θα θέλαμε να επιτύχει. Υπάρχουν λιγότερο δαπανηροί τρόποι για να επιτύχουμε όλα αυτά, ε, που δεν θα είναι και εις βάρος των φορολογουμένων και θα θέλαμε να έχουμε έναν οργανισμό ε, στον οποίο οι υπάλληλοι να μην μπορούν να απολυθούν παρά μόνο μετά από μια μακρά διαδικασία. Θέλουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα μπορεί να βοηθήσει μέσω εμπειρογνωμοσύνης, μέσω ανθρώπων όπως επισήμανε και ο κύριος Φρίξε. Παραδείγματο χάρη, εγώ θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα εξαιρετικό το γεγονό ότι το να δημιουργούμε έναν οργανισμό για να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη και τελικά Απλώς ε, δημιουργούμε ε, ένα πλαίσιο για να αναζητήσουμε πυρογνώμονες. Αν είναι να κάνουμε αυτά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πια να το κάνετε σε αυτό μόνο σας. Θα μπορούσατε ε, να το είχε κάνει η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για το μωρό, ούτε για τα νερά ε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια πολιτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτή την προσέγγιση που θα θέλαμε να ε, υποστηρίξουμε επιμένω σε εταιρική σχέση με τους εταίρους μας το χωρών και ε, θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε και όλα τα καλά στοιχεία τα οποία έχουν γίνει. Και ένα τελευταίο στοιχείο για την αποκέντρωση. Ναι, μεν αποκέντρωση, αλλά η παρούσα εμπειρία δεν μας πείθει Υπάρχει ένας έλεγχος που έχω στα χέρια μου από ένα γραφείο στην Κένια όπου διαπιστώθηκαν κάποιες παρατυπίες, ο διευθυντής παρετήθηκε. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναλάβουμε πλέον εμείς τα ενία όλη αυτή τη διαδικασία. Η ιδέα της αποκέντρωσης είναι να υπάρχει μια κάποια πυρογνωμοσύνη στα τοπικά γραφεία τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτή την οικονομική ανάπτυξη και μέσω αυτής της εμπειρογνωμοσύνης να γίνεται και ο σύνδεσμος με όλα όσα γίνονται στις Βρυξέλλες. Θεωρώ ότι υπάρχουν τα μέσα για να γίνουν όλα αυτά και ε, ε, επί της ουσίας νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Φρίξ, αλλά όσον αφορά το κέντρο ανάπτυξης επιχειρήσεων θεωρώ ότι ήγηκε η ώρα να φτάσει στο τέλος του. Ε, το γεγονός ότι θα πάψει ε, να υπάρχει δεν σημαίνει ότι θα κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει όλο αυτό ομαλά, σεβόμενοι και τα εργασιακά δικαιώματα και σεβόμενοι τους υπαλλήλους. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ε, θα ληφθεί η απόφαση τον Ιούνιο από το Κοινό Συμβούλιο Χωρώνα και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι η αρχή μιας διαδικασίας ε, phasing out, η οποία θα πάρει τουλάχιστον ε, ένα χρόνο και κατά μέγιστο δύο χρόνια. Δηλαδή θα πρέπει κάπως να ε, αναδιατυπωθεί η εντολή του κέντρου των εργαζομένων και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Θεωρούμε ότι πρέπει να επιδείξουμε και λίγο σθένος εδώ και να επιλύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεκεζέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μία πολύ σύντομη παρατήρηση. Αν ληφθεί αυτή η απόφαση που μας αναφέρετε τον Ιούνιο, μας αναπτύξατε διάφορους άξονες και μας είπατε για τη δημιουργία ενός νέου μέσου. Τότε θα ξεκινήσει και το νέο μέσο ή είναι ένα μέσο το οποίο θα είναι απλώς παροχή υπηρεσιών σε απεκεντρωμένο επίπεδο και τα υπόλοιπα θα τα διαχειρίζεστε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συστήσετε τότε κάποιο νέο οργανισμό, κάποιο νέο μέσο. Ε, με ποια σειρά θα τα κάνετε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Όλα αυτά γίνονται εκ παραλλήλου συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας, τον χωρών ΑΚΕ, για να καθορίσουμε το περιεχόμενο όλων αυτών των στοιχείων. Όπως σας είπα, το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δεν θα εξαφανιστεί τον Ιούνιο, απλώς θα ληφθεί απόφαση τον ε, Ιούνιο ε, πολιτικής και νομικής φύσεως, διότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ένα παράρτημα της Συμφωνίας Κοτονού και θα είναι μια απόφαση ε, phasing out. Επομένως, το κέντρο ανάπτυξη επιχειρήσεων θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες τους ε, για αυτό το διάστημα και φυσικά βασιζόμαστε και στη συνεργασία των μελών του κέντρου για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να ξεκινήσουμε ε, τη νέα προσέγγιση. Η νέα αυτή προσέγγιση θα είναι μια προσέγγιση η οποία θα εδράζεται στην εμπειρογνωμοσύνη και σε όλα τα στοιχεία τα οποία σας επεσήμανα, αλλά αυτή τη το κέντρο κατεβάσει τα ρολά, μου επιτρέπετε την έκφραση, τα υπόλοιπα στοιχεία, η υπόλοιπη εργαλειοθήκη θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος και πάλι στον κύριο Φρίξ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχάς να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Δεκεζέρ ποια είναι η αξία του κέντρου των επιχειρήσεων. Να σας πω το ερώτημα. Είναι ποια είναι η αξία της βασικής εντολής της αποστολής του κέντρου. Διότι αυτό είναι σημαντικό να απαντηθείτε. Μιλάμε για αντικατάσταση είτε για εξέλιξη. Το σημαντικό λοιπόν είναι να τα πάμε καλύτερα στο μέλλον γνωρίζοντας τι προϋπήρξε. Κατά την άποψή μου Ουδέποτε δεν είχαμε τόσο πολύ ανάγκη σε επίπεδο επιχειρήσεων ΑΚΕ ή νεαρών επιχειρηματιών των χωρών ΑΚΕ ή του άτυπου οικονομικού κλάδου που θα πρέπει να μπορεί να βγει από αυτή την ε, κατάσταση. Ποτέ δεν είχαμε τόσο ανάγκη από ε, εύρωστες τοπικές υποδομές που να έχουν μέσω χρηματοδότησης τη δυνατότητα πριν ε, ε, την ε, χρηματοδότηση, να στηρίξουν τις δράσεις των επιχειρηματιών ή να συνοδεύσουν τους επιχειρηματίες αυτές τις δύσκολες στιγμές της ε, πρώτης τους, των πρώτων τους κινήσεων. Αυτή είναι η εντολή, αποστολή που υπάρχει και κάποιος πρέπει να την φέρει πέρα. Το πώ είναι αντικείμενο συζήτηση και διαπραγματεύσεων. Αλλά κάπως πρέπει να γίνει. Δεύτερη προτεραιότητα επίσης είναι ότι πρέπει να διευκολυνθεί η εταιρική σχέση, οι εταιρικέ σχέσει των επιχειρήσεων, διότι στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε με την Αφρική να ε, ξυπνά πια, να ξυπνά ε, και λόγω των αναγκών που προέρχονται από την Κίνα, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και σε επίπεδο μικρομεσαίων που να παίρνουν πια διεθνή διάσταση και μέσω διαφορετικών τρόπων με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και με νέους επιχειρηματίες να βγουν και εκτός Ευρώπης. Κάποιος, κάπως πρέπει να πετύχουμε αυτές τις δύο προτεραιότητες. Εκεί θα βρεθεί η προστιθέμενη αξία που αναζητάτε. Έπειτα πρέπει να αποφύγουμε όλα αυτά να μην γίνουν με τρόπο γραφειοκρατικό, γιατί ήδη πριν από 20 χρόνια είχαμε ξεκινήσει προσπάθειες αποκέντρωσης για να πάμε την τοπική πραγματικότητα με τραπεζιτές, με συνεργασία με τους δανειοδότες μας ή τα τραπεζικά ιδρύματα, με εταιρείε ε, δημόσιας συμμετοχής μεν, αλλά στην τοπική πραγματικότητα, κοντά στους επιχειρηματίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και συγχρηματοδότηση από το επίπεδο των αντισώμενων χωρών. Και αυτό χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή ο όμιλο Ανέλ στην Αφρική, στην Ποτσουάνα, συγχρηματοδοτεί προγράμματα του δικού μας κέντρου. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους που να είναι αποτελεσματικοί και προς το κόστος και ε, προσάρμοστοι και αποτελεσματικοί. Είναι μια φυσική τάση βέβαια, δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν, αλλά θα πρέπει να ε, αναλάβουμε επιτέλους περισσότερο τα αποτελέσματα περισσότερα από τα αποτελέσματα των δύσκολων καταστάσεων, τα αίτια των δυσκολιών μας. Βεβαίως, συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Αμιλιά, ε, Βεβαίω, δεν ξέρω απλώς αν συμφωνώ με την θεωρία των τριών τετάρτων, διότι εκείνη την περίοδο το κέντρο είχε στους τομείς προτεραιότητας όπως η Αλία, η Γεωργία, ο τουρισμός, είχε προσλάβει ε, βάσει διαγωνισμού εμπειρογνώμονες πρώτου επίπεδου, τους οποίους είχαμε εξασφαλίσει έναν αριθμό ωρών εργασίας, για να έρθουν αυτοί να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες μας. Ναι, αυτό το είδος η προσέγγιση νομίζω ότι είναι αναγκαία. Αυτά θα ήταν κάποιες απαντήσεις, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ με τη συζήτηση αυτή. Η σημερινή μας συνεδρίαση λαμβάνει τέλος. Θα βρισκόμαστε αύριο με τους συντονιστές στις 9 το πρωί σε αυτή την αίθουσα και στις 10 για μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή με συγχωρείτε, Εξωτερικού Διεθνούς Εμπορίου. Θα συζητήσουμε τις εμπορικές μας συμφωνίες.